για να ακούσουμε την τροποποίηση του κανονισμού 726-2004 σχετικά με την ε, φαρμακοεπαγρύπνηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελευταία φορά εξήγησα στους αδέλφους ε, το υπόβαθρο της ε, έκθεσης περί φαρμακο επαγρύπνησης ε, και η όλη υπόθεση ξεκίνησε με ένα φάρμακο που κυκλοφορούσε σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και κάπου αλλού για τον διαβήτη ε, Και προέκυψαν διάφορα ζητήματα και σιγά σιγά η εταιρεία το απέσυρε από τις διάφορες αγορές ε, πλην της Γαλλίας. Όταν όμως προέκυψε η υπόθεση και ήταν μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και ακόμα υπάρχει, υπάρχουν υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια, η Κομισιόν επανεξέτασε την νομοθεσία φαρμακοεπαγρύπνησης που είχαμε εγκρίνει πριν από 18 μήνες και παρά το ότι πολλά πράγματα γίνονται πιο αυστηρά, η Κομισιόν βρήκε κάποια πιθανά παραθυράκια τα οποία δικηγόροι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Δεν θα το έκαναν οι περισσότερες εταιρείε, αλλά στην περίπτωση της Σερβιέ αυτό το οποίο συνέβη είναι πως ε, όταν αντιμετώπιζε προβλήματα το απέσυρε ε, όχι για λόγους ασφαλείας, δεν ζήτησε καν άδεια στην Ισπανία και την ε, Ιταλία. Οπότε η νομοθεσία μας δεν καλύπτει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή τι γίνεται όταν μια εταιρεία αποσύρει ένα φάρμακο από την αγορά εθελοντικά. Καλύπτει τα προβλήματα ασφαλείας λοιπά. Οπότε η Κομισιόν εδώ πέρα κατέθεσε κάποιες αλλαγές για να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια. Και βεβαίως Είχαμε συναντηθεί οι ισχυώδεις εισηγητές για την ανάγκη να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια. Κοιτάξτε, η νομοθεσία αυτή θα τεθεί ενισχύ τον Ιούλιο και αυτό το οποίο ελπίζουμε εγώ ως εισηγήτρια και οι εισηγητές και το Συμβούλιο και Κομισιόν είναι να συμφωνήσουμε γρήγορα για να εφαρμοστεί η νομοθεσία όλοι μαζί γιατί έτσι θα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές ε, και εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στο Λονδίνο που έχει ενισχυμένο ρόλο να ε, εφαρμόσουν τώρα ένα μπλοκ νομοθεσίας και να προετοιμαστούν σωστά. Και είναι σημαντικό και για την ασφάλεια των ασθενών να κλείσουμε τυχόν παρατηράκια. Οπότε, Κομισιόν δεν θα αναφέρω τώρα όλες τις προτάσεις της. Ε, κάνει τέσσερις αλλαγές. Εάν μια εταιρεία αποφασίσει να μην ανανεώσει μια άδεια, πρέπει να δηλώσει γιατί το κάνει αυτό. Πρέπει να το πει στη ρυθμιστική αρχή. Οπότε οι ε, εταιρείε θα συμπεριφέρονται με τρόπο διάφανο. Εάν αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας, θα ξεκινήσει μια διαδικασία αυτομάτως εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Στο παρελθόν ήταν στη διακριτική ευχέρεια των, κρατών μελών. Και βεβαίως στην περίπτωση του Σεργέ είχαμε πρόβλημα. Και τέλος, το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό της επιπρόσθετης ε, παρακολούθησης των φαρμάκων αν κάποιο είναι π.χ. νέο φάρμακο, για πέντε χρόνια το παρακολουθούν οι ιατροί και οι λοιποί. Και τους λένε να αναφέρουν τις παρενέργειες. Στη νέα μας νομοθεσία θα το ξέρουν και οι ασθενείς. Θα υπάρχει ένα μαύρο τρίγωνο που θα σημαίνει νέο φάρμακο και σημαίνει πρέπει να μας βοηθήσετε, εμάς, τους γιατρούς, αν υπάρχουν προβλήματα να μας τα πείτε. Αλλά Υπάρχει και συμπληρωματική ε, παρακολούθηση, η οποία όμως δεν κάλυπτε τις ε, περιπτώσεις μιας μελέτης ασφαλείας μετά την αδειοδότηση. Γιατί συχνά λένε εντάξει μπορείτε να το βγάλετε στην αγορά αλλά κάποια πράγματα ακόμα πρέπει να τα δούμε και να γίνει μια μελέτη. Στην περίπτωση του Mediator ε, είχε ζητηθεί μια τέτοια μελέτη κάπου γύρω στο 2001 και ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε το 2009 πριν αποσυρθεί από την αγορά. Είναι δυνατόν οι εταιρείε να μην κάνουν αυτές τις μελέτες και πρέπει να φροντίσουμε η επιπλέον παρακολούθηση να συμβαίνει μέχρι να τελειώσουν οι μελέτες και τότε μπορεί να βγει από τη λίστα το φάρμακο. Αυτά είναι τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν. Η έκθεσή μου στηρίζει σε γενικές γραμμές τις προτάσεις της Κομισιόν. Θέλω να φροντίσουμε εδώ πέρα το να είναι εδώ πέρα τα πράγματα ξεκάθαρα και πρέπει να βρούμε μια διατύπωση, γιατί η Σερβία είχε πει είναι για εμπορικού λόγου και το αποσύρουμε από την Ισπανία και την Ιταλία. Τώρα εξετάζει και το Συμβούλιο αυτό το ζήτημα και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με το Συμβούλιο. Ήδη τους έχουμε μεταφέρει τις ανησυχίες μου για κάποιες αλλαγές που έκαναν στην πρόταση της Κομισιόν και συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ καλά. Το νέο σχέδιο του Συμβουλίου είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μου τροπολογίες και, τις, ε, και την πρόταση της Κομισιόν. Ζητάω λοιπόν από τους συναδέλφους να ελεξιτοποιήσουμε τις ε, τροπολογίες γιατί αν έχουμε πολλές ε, τροπολογίες θα πάει η εφαρμογή πέρα από τα μέσα Ιουλίου. Τώρα υπάρχει μια τροπολογία που σκέφτονται να καταθέσουν οι συνάδελφοι. δεν είναι εδώ βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντική. Μια τροπολογία λοιπόν για αυτό το οποίο λέμε μια χρήση ε, εκτός από την ενδεικνυόμενη. Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρουν οι οδηγίες. Γιατί αυτό ήταν φάρμακο για το διαβήτη και το έπαιρναν για να δυνατήσουν. Οπότε θα περιοριστεί αυτή η χρήση και υπάρχουν ειδικοί κανόνε για αυτέ τι περιπτώσει, Αλλά να πω το εξή ε, είναι κάτι το πολύ πολύπλοκο. Γιατί πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να πει στο γιατρό πώ θα γράψει το φάρμακο. Οι γιατροί είναι ελεύθεροι να λάβουν την απόφαση αυτή. Και όταν συζητούσαμε για τα παιδιατρικά φάρμακα, το λέμε πολλέ φορέ. Σε πολλέ περιπτώσει για τα παιδιά τα γράφουν για άλλε χρήσει και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχει και σοβαρό, σοβαρά εμπορικά συμφέροντα γύρω από αυτό το ζήτημα. Παραδείγματος χάρη στη χώρα μου. Έχω κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις, αλλά στις ειδήσει τρίτη πρωί άκουσα πως στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποια υγειονομικά συστήματα χρησιμοποιούν ένα φάρμακο ε, κατά του καρκίνου για κάποιες ε, εκφυλιστικές ε, ασθένειες των ματιών που είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Και φαίνεται πως λειτουργεί. Οι γιατροί θεωρούν πως λειτουργεί. Αλλά τώρα η Νοβάρτης πήγε στο δικαστήριο να σταματήσει το, για να σταματήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να το χρησιμοποιεί για άλλη χρήση. Τώρα δεν έχω δει τις λεπτομέρειες, μόνο τον τύπο. Αλλά δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να αποφασίζει η φαρμακευτική εταιρεία τι μπορούν να συνταγογραφήσουν οι γιατροί και τι μπορεί να δώσει το σύστημα υγείας. Είναι περίπλοκο το ζήτημα και δεν θέλω να αποφασίσουμε εμείς το πώ θα ρυθμιστεί αυτή η χρήση. Χαίρομαι που έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Και το συζητάμε με Συμβούλη και Κομισιόν, αλλά αν αρχίσουμε να καταθέτουμε τροπολογίες για αυτό το θέμα τώρα, δεν θα τελειώσουμε τον Ιούλιο, ούτε καν τον επόμενο Ιούλιο. Γιατί είναι δύσκολο το ζήτημα. Τα συμφέροντα είναι μεγάλα, όπως σας είπα, αφορούν ευρεσιτεχνίες κτλ. Οπότε προτιμώ οι συνάδελφοι να σκεφτούν πάρα πολύ προσεκτικά το ζήτημα. Αλλά λείπουν τώρα αυτοί που θέλουν να καταθέσουν τις τροπολογίες, θα τους γράψω ένα σημείωμα. Είναι λοιπόν πολύ σύντομη προθεσμία για τις τροπολογίες. Ελπίζουμε να μην έχουμε τροπολογίες ή ελάχιστες και να πάμε γρήγορα σε ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε να με το Συμβούλιο που αντιδρά πολύ καλά και γρήγορα να έχουμε ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Αγιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μακάβαν γιατί έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Ε, μια μεγάλη δουλειά. Και Συνεδρίασε με τους κοιόδης εισηγητές, όπως ακριβώς είχαμε συμφωνήσει. Και επίσης, συμφωνώ ότι δεν πρόκειται για μια νέα νομοθεσία. Θέλουμε να αναθεωρήσουμε μια παλιά νομοθεσία λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με την υπόθεση του mediator. Και με την υπόθεση των ε, stress test. Ελπίζω να μπορέσουμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε αυτό το πρόβλημα αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να λύσουμε όλα τα προβλήματα που σας ανέφερε η Λίντα. Αυτό είναι αδύνατον. Είναι, κάποια θέματα είναι ευθύνη των γιατρών και των υγειονομικών αρχών. Το πώς θα χρησιμοποιήσουν κάποια φάρμακα. Δεν μπορούμε, όποια νομοθεσία του κόσμου και να έχουμε, να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Συμφωνώ με την έκθεσή της, με τις τροπολογίες που είναι πολύ συγκεκριμένες, έτσι για να ρυθμίσει κάποια συγκεκριμένα σημεία της πρότασης της Κομισιόν που γενικά είναι καλή, όπως η τροπολογία 3 που μιλάει για την υποχρέωση των κατόχων να έχουν άδεια εμπορίας και που είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση που θέλουν να μην ανανεωθεί αυτή η άδεια να ενημερώσουν τα κράτη-μέλη. Γιατί, ας πούμε, στην υπόθεση του mediator είπαν ότι δεν θέλαν να ανανεώσουν αυτή την άδεια γιατί δεν υπήρχε ζήτηση. Ενώ το πρόβλημα στην πραγματικότητα από πίσω ήταν άλλο. Κρυβόταν κάτι πολύ μεγάλο από πίσω. Θέλω να ρωτήσω τώρα την Κομισιόν. Σε περίπτωση της ε, διαδικασίας του κατεπήγοντος. Σε αυτό το άρθρο που μιλάτε για αυτή τη διαδικασία. Όταν υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας λέτε ότι θα πρέπει να ε, καταφύγουμε σε αυτή τη διαδικασία κατεπήγοντος και θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση μέσα σε 60 μέρες ε, από την ε, υπηρεσία φαρμάκων. Μήπως έτσι βαραίνουμε πολύ την υπηρεσία φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τελεσπών Φαρμάκων, ο οποίος έχει πάρα πολλή δουλειά ήδη. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μου απαντήσει. Με βάση τις πληροφορίες που έχει, ο οργανισμός μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Επίσης, ε, θέλω να συστήσω και εγώ να μην υποβάλλετε πάρα πολλές τροπολογίες. Το βασικό είναι να μπει ε, σε εφαρμογή αυτή η νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην υποβάλλετε τροπολογίες πέραν των απολύτως αναγκαίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατόπιν έχουμε την κυρία Γερακουδάκη. Έχετε το λόγο. Να σας το πω ταχαίως για να συμφωνήσω με τον εισηγητή. Την εισηγήτρια, εν πάση περιπτώσει, αν θα γίνουμε αυτά τα παραθυράκια και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσέγγιση της βασικής νομοθεσίας. Ε, εδώ και καιρό προετοιμαζόμαστε, κάποια στιγμή το να έχουμε ολοκληρώσει και επομένως και η δική μας πολιτική ομάδα θα υποστηρίξει την εισηγήτρια και ελπίζουμε ότι θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεση ταχαίως από την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Ροτ για τη χρήση που δεν αναφέρονται στις ε, οδηγίες χρήσης. Ε, με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες ε, είναι υποχρεωμένες να γράφουν για ποιο λόγο χορηγείται αυτό το φάρμακο και για ποιο επίσης ασθένειες κτλ. Μπορεί αν εμείς τώρα επιτρέψουμε και άλλες χρήσεις να δημιουργηθεί πρόβλημα. Εγώ θέλω να υποβάλω μόνο μία τροπολογία. Το έχω πει ήδη στην εισηγήτρια. Ε, καταρχάς, ε, ευγνώμων προς την εισηγήτρια. Ε, οι τροπολογίες που έχει προτείνει η εισηγήτρια είναι πολύ καλές. Παραδείγματο χάρη, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κενά και παραθυράκια σε μια νομοθεσία αμέσω, να προτείνουμε να τα καλύπτουμε. Και επίση, ε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που πει η εισηγήτρια ότι όταν φεύγει κάτι από την αγορά, να ξέρουμε γιατί φεύγει από την αγορά. Ε, κάτι που ξέχασε όμως η Κομισιόν. Γι' αυτό στράφαμε προς την Κομισιόν. Το θέμα των τελών. Δεν υπάρχει καν κανονισμός για τα τέλη. Στην ε, τελευταία, στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φαρμάκων ακούστηκαν πολλές επικρίσεις για το γεγονός ότι πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά η ΕΜΑ, αλλά δεν έχει καμία ιδέα για το τι πρέπει να κάνει για τα τέλη. Ε, βρίσκομαι μεταξύ Σκύλας και Χάριφης τώρα. Ε, μήπως πρέπει να έχουμε ένα καονισμό για τα τέλη, αλλά αν το κάνουμε στην απόφαση θέλουμε ε, ένα μισή χρόνο, το λιγότερο, ή δύο χρόνια. Ε, η άλλη λύση είναι μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εφόσον, να το δεχτούμε αυτό, εφόσον μπορούμε να εμπιστευτούμε την Κομισιόν. Αν η Κομισιόν προχωρήσει ε, το θέμα των τελών μέσω κατεξιοδότηση πράξης, να την υποστηρίξω την Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν φαίνεται λίγο ανήσυχος. Θα θέλαμε κάποια εφαρμοστική νομοθεσία για τα τέλη. Και ελπίζω να έχω την υποστήριξη και της συγγήτρια και των υπολείπων. Ευχαριστώ. Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Λίντα. Συμφωνώ με την Πιλάρ Αγίζο πως είναι πολύ καλή αυτή η δουλειά. Συμφωνώ και με τη Λίντα και την Πιλάρ πως πρέπει να είμαστε προσεκτική για το θέμα της χρήσης εκτός ε, των οδηγιών. Ένα νέο θέμα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά σε τόσο λίγο χρόνο. Δεύτερον, είναι σωστό πολιτικά να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε αυτή τη χρήση. Γι' αυτό αυτό κάναμε π.χ. και στα παιδικά φάρμακα. Αλλά χοντρικά θα εκτιμούσα θυμάστε και την έκθεση Φρανσουάζ Κροστέτ ε, καταφέραμε στην ε, στις μονάδες εντατικής θεραπείας να μειωθεί η περίπτωση από το, η χρήση από το 90% στο 80% και είναι Ηράκλειο το έργο του να κατέβει κάτω από εκεί. Και τι είναι δεν θέλουμε να μην έχουν τα παιδιά τα φάρμακα που χρειάζονται για να ζήσουν, γιατί δεν έχουν ε, την ε, άδεια τα φάρμακα. Μπορούμε λοιπόν να το μειώσουμε, αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπεται καν νομικά να δυσκολέψουμε αυτή τη χρήση. Πρέπει να το, να το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά με την Κομισιόν. Αλλά όχι σε αυτή την έκθεση. Οπωσδήποτε όχι. Έχω κάτι ακόμα να πω. Δεν θέλω να περιπλέξω τη διαδικασία, αλλά υπάρχει κάτι που είχε μείνει από την αρχική χρήση του 2010. Το κουτί με τις πληροφορίες ε, του φαρμάκου η Κομισιόν είχε προτείνει μια σύνοψη των σημαντικότερων ιδιωτήτων του φαρμάκου στη συσκευασία. Και η Επιτροπή το υιοθέτησε. Δεν υπήρξε έτοιμα διαγραφής. Μετά πήγε η Λίντα στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν το δέχτηκε. Δεν ξέρω, ίσως να μην έδωσαν ιδιαίτερο οι ομάδες. Μας το λένε ξανά ανεξάρτητοι ειδικοί πως είναι καλό αυτό το σύστημα για να βελτιωθεί και η φαρμακοεπαγρύπνηση, οπότε στην Ολομέλεια, πάνω από την Επιτροπή μας δηλαδή, υιοθετήσαμε στην έκθεση Φιέλνερ μια σχετική τροπολογία. Δεν θέλω λοιπόν να το θάψουμε αυτό το θέμα. Αντίθετα πρέπει να δώσουμε μια οδηγία προς την Κομισιόν για το ότι θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό έχω μία τροπολογία. Ευχαρίστως να την αποσύρω, εάν συνεννοηθούμε πως είμαστε υπέρ και σε κάποια άλλη στιγμή θα το δούμε σοβαρά. Κάποια στιγμή, αν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα με το Συμβούλιο σε μια άλλη νομοθετική διαδικασία. Για... Ζητάω κατανόηση, σας το είχαμε αποφασίσει στην Ολομέλεια και μέσω αυτής της ε, ευτυχούς ε, διαδικασίας εξαφανίστηκε. Γι' αυτό ήθελα να το υπενθυμίσω και θα καταθέσω και σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ. Τη σχεδόν των φιλελευθέρων, η κυρία Παρβάνοβα. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για το σχέδιο της έκθεσης και για την άρεστη συνεργασία που είχε η συγγήτρια με τους σκιώδες συγγητές. Έτσι τα πράγματα γίνανε ευκολότερα και έτσι θα ενημερώσουμε αυτό το σημαντικό νομοθέτημα. Η Επιτροπή επίσης θα συμβάλλει κατόπιν του ότι επισημάθηκαν αυτά τα κενά, τα παραθυράκια και είχαμε και το θέμα του διαμεσολαβητή του Γάλλου και θα καλυφθεί και η πρόταση της Λίντα. Αυτό με την ενεργοποίηση της διαδικασίας του κατεπήγοντος όταν προτίθεται κάποιος να αποσύρει ένα προϊόν για λόγους ασφαλείας, όπως έγινε με τον Ιεμισοδευτή σε διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαστε να έχουμε επιπλέον εποπτεία και είμαστε επίσης υπέρ του να υπάρχει αιτήσια δημοσίευση για τα προϊόντα για τα οποία ανακλήθηκε η έγκριση κυκλοφορίας και αυτό να είναι αιτιολογημένο. Επίσης, συμφωνώ με την πρόταση που τώρα συζητούμε. Πιέζει ο χρόνος σε σχέση με τη Συμφωνία του 2010 και γι' αυτό είναι σημαντικό να αντιδράσουμε στις πρόταση της Κομισιόν και να εστιάσουμε την προσοχή μας στο στόχο που έχουμε τάξει όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας. Όσον αφορά τώρα τη χρήση των φαρμάκων αυτών, είναι αλήθεια ότι είπε ο για τη χρήση εκτός ετικέτας και για τα τις έγκρισης για τέτοιες πρακτικές. Οπότε και αυτό θα καλυφθεί από την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Δεν έχουμε και τώρα φρέσκες εξελίξει σχετικά σχέση με την Οβάρτη στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό να μελετηθεί, να ληφθεί υπόψη και να είμαστε προσεκτικοί για κάποιε τροπολογίε. Του έριξα μια ματιά και να μην ξεχνούμε τη διάταξη του άρθρου 5 που λέει για τις εξαιρετικές περιστάσεις όσον αφορά τα μη εγκεκριμένα προϊόντα και την ευθύνη του τους Και να δούμε τι θα γίνει για τον ασθενή όσον αφορά τη χρήση εκτός της ετικέτας. Προσοχή, προσοχή σε αυτό το σημείο και ίσως θα πρέπει ε, ο Οργανισμός για τα Φάρμακα, η Υπηρεσία για τα Φάρμακα, κοινοτική, να προσέξει την σωστή εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας των Καταναλωτών. Έχετε τον λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να απαντήσω στα διάφορα σχόλια. Υποστηρι... Ε, σημειώνω την υποστήριξη προς την πρόταση της Κομισιόν. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τους λόγους που μας ε, ανάγκασαν να υποβάλουμε την ε, πρόταση. Σας ευχαριστώ για αυτό, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Η κυρία Γιούζο ζήτησε αν η διαδικασία κατεπήγοντος θα καλύψει και την αλλαγή ενδείξεων κτλ. Ναι, αυτό έχει προβλέψει η Κομισιόν. Ήταν σημαντικό αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει όταν τίθεται θέμα, σοβαρό θέμα ασφάλειας σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα του φαρμάκου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κομισιόν. Δεύτερο σημείο ε, της κυρίας Ροτμπέρεν, το θέμα των τελών. Σας διαβεβαιώ ότι ε, είμαστε σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Φαρμάκων και σήμερα ακόμα θα ξεκινήσουμε μια διήμερη συνάντηση με τα μέλη του προσωπικού της, του οργανισμού αυτού, ούτως ώστε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα των τελών και να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα το υποβάλουμε στους ενδιαφερόμενους φορείς, στους stakeholders, για να γίνει μια δημόσια διαβούλευση. Και, εν συνεχεία, με βάση αυτό θα υποβάλουμε την πρότασή μας. Τώρα, αν χρειαστεί σοβαρή και πλήρης και 100% συναπόφαση, στην καλύτερη περίπτωση θα χρειαστούμε ένα χρόνο. Ε, δεν σταθεί κανένας γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν διάφορα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν και διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν ένα χρόνο, αλλά πάντως ε, το... είμαστε σε άμεση επαφή με την ε, αίμα, τον οργανισμό φαρμάκων για αυτό το θέμα. Εν συνεχεία, έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη για το θέμα των ιδιωτήτων του φαρμάκου και για το φυλάδιο με τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνει η συσκευασία. Και θέλουμε να δούμε τι στοιχεία αναφέρει το, η συσκευασία Ξέρετε ότι ε, αυτές οι πληροφορίες που δίδονται πάνω στο κουτί του φαρμάκου ε, είναι κάτι που το ξεκίνησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια, ξεκινάμε μια μελέτη για να δούμε τι πρέπει να γίνει για να είναι πιο ευανάγνωστες αυτές οι οδηγίες πάνω στο κουτί και να λάβουμε υπόψη ε, τι υπάρχει πάνω στο κουτί και στις οδηγίες χρήσης. Τώρα, για τη χρήση του φαρμάκου πέρα από αυτά που αναφέρουν οι οδηγίες. Είναι κάτι περίπλοκο, όπως υπόθηκε και θα χρειαστεί να το σκεφτούμε πολύ πιο ενδελεχώς πριν, το... πριν προτείνουμε οτιδήποτε. Άκουσα διάφορες ανησυχίες που εκφράστηκαν για τον κανονισμό τέτοιας χρήσης φαρμάκων, που ασχολείται με τέτοια χρήση φαρμάκων. αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγο έχει το Συμβούλιο, γιατί ζήτησε το λόγο και για την Προεδρία του Συμβουλίου θα ακούσουμε την κυρία Πάουλσον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που είμαι ενώπιόν σας σήμερα για να συζητήσουμε την πρόταση αυτή για τη φάρμακο επαγρύπνηση. Είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου που ασχολείται με θέματα υγείας. Είμαι νομικός και έχω ασχοληθεί με θέματα υγείας στο Υπουργείο Υγείας της Δανίας. Χαίρομαι που γίνεται λόγος για το θέμα αυτό και ελπίζω οι νέοι κανόνες να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω ότι μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα πως το θέλει όλο το Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αποφασίσαμε τρεις αλλαγές. Η πρώτη αφορά την διαδικασία της Ένωσης για το άρθρο 117 ε. η Επιτροπή με την, τι γίνεται με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, τι αρμοδιότητες έχουν, πώς λαμβάνονται οι γρήγορες αποφάσεις και δεν θεωρούμε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να βουλιάξει κάτω από υπερβολικές αρμοδιότητες, γιατί έχει ήδη αρκετές. Αρκετές και δύσκολες μετά από την νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2010. Γι' αυτό λοιπόν εκφράζουμε την ευχή οι διαδικασίες της Ένωσης να μην οδηγήσουν ε, σε δρομολόγηση πολλών διαδικασιών αυτόματων. Επίσης, υπάρχει το άρθρο 23 του κανονισμού που αφορά το λεγόμενο μαύρο σύμβολο. Με βάση την αξιολόγηση του Συμβουλίου, αυτό το μέτρο μας φαίνεται πολύ ευρύ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το σημείο, να το αξιολογήσουμε. Γιατί Μόνο όταν υπάρχει σοβαρότατη και εντονότατη ανησυχία θα πρέπει να αποδίδουμε αυτό το σύμβολο. Και οι χρήστες των φαρμάκων, οι ασθενείς, θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα γιατί α, μπαίνει αυτό το μαύρο σύμβολο. Γιατί αυτό υπήρχαν προβλήματα από την αρχή ή προέκυψαν νέα στοιχεία. Ούτως ή άλλως πρόκειται για προϊόντα που έχουν άδεια εμπορίας. Μην το ξεχνάμε. Τα φάρμακα αυτά έχουν την άδεια αυτή. Επομένως θα πρέπει να μην υπάρξει καμία σύγχυση στο μυαλό του ασθενούς. Επίσης, άρθρο 123 της οδηγίας. Διατάξει σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Τις δίδουν οι αρχές για την περίπτωση που τίθεται στην εμπορία νέα προϊόντα ή στην περίπτωση που ένα προϊόν, φάρμακο δηλαδή, ζητάει ανανέωση της άδειας. Αυτός ο κύκλος πληροφόρησης θα πρέπει να κλείνει ούτως ώστε και τα κράτη-μέλη στα οποία δεν υπάρχει εμπορία αυτού του συγκεκριμένου φαρμάκου να ενημερώνονται ε, για το τι συμβαίνουν σε άλλες αγορές. Για να υπάρχει ασφάλεια στο επίπεδο το ιατρικό. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πληροφορίες πολύ σημαντικές γιατί ακριβώς αφορούν την ασφάλεια της υγείας. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης στο Συμβούλιο, ασχοληθήκαμε με την περίπτωση μιας άδειας σε τρίτες χώρες για προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν γι' αυτό. Για να κλείσω, θέλω να επαναλάβω ότι η Δανέζικη Προεδρία, εν ονόματι του Συμβουλίου, είναι έτοιμη να δρομολογήσει έναν επικοδομητικό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για αυτές τις δύο προτάσεις. Ευχαριστώ. Θα δώσω ξανά το λόγο στην Ελίνα Μακάβνη για να κλείσουμε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για την στήριξή τους. Ε, άκουσα πως θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες. είμαι σίγουρη πως θα τις δούμε. Για τη χρήση τώρα τιμή ενδεικνυόμενη καλό είναι οι συνάδελφοι να αναλάβουν μια ξεχωριστή πρωτοβουλία γιατί είναι πολύ πολύ πολύπλοκο το θέμα. Ίσως πρέπει να γίνει μια ακρόαση και να το σκεφτούμε. Τι κατευθυντήρε γραμμέ του οργανισμού φαρμάκων κτλ. Αλλά πριν ε, μπει μέσα, Αντωνία, εγώ μίλησα για του γιατρού που τα γράφουν και το ότι αυτοί είναι αρμόδιοι. Δεν μπορούμε να το λύσουμε έτσι εύκολα. Γι' αυτό το οποίο είπε η κυρία Γιούζο για την αίμα και το, την επιβάρυνσή της. Πρέπει να φροντίσουμε να δουλεύει. Δεν είναι πλέον μια αίθουσα συνεδριάσεων στο Λονδίνο όπου κάποιοι μαζεύονται και μιλάνε. για τις ανησυχίες τους για τα φάρμακα. Οπότε νομίζω πως ε, η περίπτωση με διατόρο δεν θα επαναληφθεί. Αυτό πρέπει να, να αλλάξει. Και καθώς μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, εγώ έχω ήδη νούμερα για το πόσες περιπτώσεις απασχολούν το χρόνο την ε, υπηρεσία φαρμάκων. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να φροντίσουμε. Το ένα είναι το κατεπήγον, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει επίσης να εξετάσουμε και είναι άλλη αυτή η διαδικασία. Στο άρθρο 31 αυτό το οποίο συνέβη με το Mediator είναι πως το συζήτησαν πολλές φορές στην υπηρεσία. Φαίνεται αυτό στα πρακτικά, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να μαζεύονται και να μιλάνε. Τώρα, αν τους πληρώνουμε, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ευθύνες και να λαμβάνουν αποφάσεις. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να βρούμε μια λύση. Αν υπάρχουν πραγματικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο ένα ή στο άλλο επίπεδο. Και αν όχι πρέπει να ξέρουμε γιατί. Νομίζω λοιπόν πως το σύστημα πρέπει να συμμαζευτεί. Ξέρω πως όλες οι ρυθμιστικές αρχές ε, θέλουν να το κάνουν αυτό. Ανησυχούν για την περίπτωση Mediator. Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι. Ελπίζω να συμφωνήσουμε έτσι ώστε μέσα Ιουλίου να έχουμε πολύ καλύτερη ασφάλεια ε, των φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όσου μίλησαν. Ευχαριστώ την Προεδρία που ήρθε στην Επιτροπή μας. Η προθεσμία για α, τις ε, τροπολογίες είναι 27 Απριλίου και συμφωνήσαμε με την εισηγήτρια για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα γιατί ψηφίζουμε το Μάιο, 8 Μαΐου όλες οι τροπολογίες μπορούν να καταστούν μόνο στα αγγλικά και να ψηφίσουμε την έκθεση το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Και βεβαίως η γραμματεία μου λέει εδώ πέρα πως ευχαρίστως είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει στην διατύπωση των τροπολογιών στα αγγλικά. Ωραία, περνάμε στο σημείο 20 της μερική διάταξης, το οποίο είναι εθελοντική και μη αμοιβόμενη δωρεά ιστών και κιτάρων. Εδώ πέρα η συγγήτρια είναι η κυρία Η κυρία Γιανακουδάκη. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Και ευχαριστώ τους κοιόδες συγητές με του οποίου σήμερα συναντήθηκα. Ακούγομαι, ναι. Διότι με βοήθησαν πάρα πολύ και η λέξη κλειδί σε αυτή την έκθεση είναι εθελοντική και γι' αυτό και λέμε να υπάρχει τέτοια αγνευσιμότητα και διαφάνεια σε σχέση και με την έκθεση που έχουμε κάνει στις αρχές της χρονιάς όσον αφορά τις δωρεές οργάνων. Δηλαδή, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να δίνει εθελοντικά και δωρεάν τέτοια κύτταρα, αίμα, βλαστοκύτταρα κλπ. Πάρα πολύ χρήσιμο θα είναι αυτό και πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι αυτά σώζουν ζωές. Ομφαλοπλακουντικό αίμα και επίσης να έχουμε συμμετοχή ιδιωτικών και δημοσίων κρατικών νοσοκομείων. Καλά κρατικές αλλά θα πρέπει backup να έχουμε τις ιδιωτικές και να συνεργάζονται και ιδιωτικέ τράπεζε. αίματο. Αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμο είναι ότι έχουμε κάτι το οποίο ονομάζεται ε, μία αμοιβόμενη βάση. Δηλαδή, εδώ κάποιοι να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιες ιατρικές αγωγές και θεραπείες εύκολα και οπότε έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στην, αύξηση των δωρεών, οαρίων, σπέρματος κλπ. Και γαμετών. Και να σας τα πω με δύο λόγια. Στην περίπτωση της δωρεάς οαρίαν μπορεί κάποια γυναίκα να δωρήσει κάποια οάρια και ταυτόχρονα κάνει και τη δική της θεραπεία για την ε, τεχνητή γονιμοποίηση, την vitro, και Αυτό μειώνει την αμοιβή που να πληρώσει την κλινική και υποφελεί και κάποιον άλλο. Το ίδιο ισχύει για το σπέρμα και για την κατάψυξη που προβλέπεται. Δηλαδή, για κάποιες θεραπείες μελλοντικές, 3-5 χρόνια, καταψύχουν τα οάρια, εάν το δωρήσει άλλα οάρια. Και έτσι, διευκολύνεται η πρόσβαση για περισσότερους οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα ενδεχομένω. Η προθεσμία της τροπολογίας είναι νομίζω τρεις του μηνός, αν θυμάμαι καλά. Ναι, τρεις. Και σε αυτή τη φάση, παρακαλώ, πέστε μου τη γνώμη σας και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Περνάμε σκιώδης. Ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Μαρίνα για να κουτάκι για τη δουλειά που έχει κάνει. Πραγματικά είναι πολύ καλή βάση για τη δουλειά μας στο σχέδιο έκθεση. Έχει ένα σαφές μήνυμα. Θέλουμε οι δωρητές ε, ιστού και οργάνων να δωρίζουν χωρίς ε, αμοιβή. Επίσης υποστηρίζω το σημείο 23 απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει δηλαδή μια σαφής ε, νομική ρύθμιση για τους ε, δωρητές κάτι το οποίο βέβαια δεν ήταν τότε όταν πέρασε η οδηγία δυνατόν να συμβεί δεν το ήθελε Συμβούλιο και Κομισιόν αλλά οι καιροί αλλάζουν η Μαρίνα Γιανακουδάκη αναφέρεται στην οδηγία περί ε, δωρητών οργάνων όπου έχουμε έχουμε πει με συμφωνία Κομισιών και Συμβουλίου πως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να είναι εθελοντικοί και ε, χωρίς αμοιβή η προσφορά αυτή. Και ο λόγος είναι πως τότε ήταν διαφορετική η νομική κατάσταση όταν ευθύθηκε η οδηγία. Εν τω μεταξύ υπάρχει η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας πως η μη εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος είναι πλέον αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Γι' αυτό αυτό το οποίο αναφέρεται στο 23 είναι πάρα πολύ έξυπνο, ζητάμε δηλαδή από την Κομισιόν να προσαρμόσει αυτές τις διατυπώσεις και στο επίπεδο της οδηγίας ε, προσφοράς ε, οργάνων είναι βασικό για εμένα. Η λασιμότητα επίσης σημαντικό και στο σημείο 9 μιλάμε για το ζήτημα του εμπορίου στο διαδίκτυο με τους ε, γαμέτες. Επίσης για το αίμα του ομφάλιου λόρου. Νομίζω πως αναφέρεται εδώ πέρα πως ε, τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν πως η δωρεά είναι ε, εθελοντική και τα Νομίζω πως ισχύει αυτό οπωσδήποτε και για το αίμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Σωστό είναι αυτό λοιπόν το οποίο έχει κάνει εδώ πέρα η Μαρίνα για να κουδάκι και το θέτει στο προσκήνιο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις ιδιωτικές αυτές ε, τράπεζες αίματος ε, του Μιχαήλου και αν θα τις εξισώσουμε με τις ε, δημόσιες. Ε, ούτως ή άλλως ε, έχει προχωρήσει η επιστήμη και ξέρουμε τώρα πολύ περισσότερο τι θεραπείες μπορούν να γίνουν και είναι ηθικά το καλύτερο αυτό, αλλά δεν πρέπει και τις ιδιωτικές τράπεζες να τις απαγορεύσουμε ή να, την, να τις φέρουμε σε δυσχερέστερη θέση. Αν τηρούν ε, τις προδιαγραφές ασφαλείας ε, κτλ. Και την αρχή βεβαίως του ότι δεν υπάρχει εμπορευματοποίηση με κύτταρα και ιστούς όπως αναφέρεται στη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, το εγγυώνται αυτό και οι ιδιωτικέ αυτές τράπεζες έχουν το ρόλο τους και ε, πρέπει να ξεκαθαρίσει άρα ποιες δυνατότητες υπάρχουν για θεραπεία και ποιες δεν υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να βελτιωθεί σε κάποια σημεία η έκθεση γιατί η φυστάμενη νομοθεσία δεν είναι τέλεια αλλά νομίζω πως μπορούμε να πείσουμε την ψυχή να τη δει λίγο κάπως. Ο εκεί που λέει στην οδηγία στα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ε, προσφορά, να, την εθελοντική και μετά στις αιτιολογικές σκέψεις παρόλα αυτά στο ΆΕ διαβάζουμε πως ε, κάποιες χώρες έχουν λάβει μέτρα στόχος των οποίων είναι η αυτάρκεια σε ιστούς και αίμα και όργανα νομίζω πως δεν ε, ταιριάζει αυτό ούτως ή όλες μόνο 11 κράτη-μέλη ε, ε, έχουν κάνει τέτοιες προσπάθειες. Επίσης, Πριν από χρόνια είχαμε την ε, συζήτηση για τους δωρητές από τη Ρουμανία που τους πλήρωναν τους μισθούς ενός εξαμήνου για να δωρήσουν όργανα και κινδύνευε η ζωή τους. Ε, δηλαδή, μισθή έξι μηνών τι... Και είναι και εμπορευματοποίηση, είναι ντροπή. Ε, εδώ πέρα ε, έχουν δείξει συνάδελφοι οπωσδήποτε από την Δανία που έρευσαν τα χρήματα. Πρέπει να πούμε πως δεν αποδεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις και μπορούμε να κάνουμε κάτι στο πλαίσιο της ε, νομοθεσίας και να γίνει αυστηρότερη. Και τέλος, η Μαρίνα ανέφερε την πληρωμή σε είδος. Εδώ πρέπει να το δούμε αυτό. Εάν ε, το θέμα είναι ότι ένα ζευγάρι δεν είναι σε θέση γιατί υπάρχει μια ξέρω η γυναίκα είναι άρρωστη και δεν μπορεί να κάνει παιδιά και σε, άλλη, σε ένα άλλο ζευγάρι δεν έχει ο άντρας σπέρμα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε. Αν όμω μιλάμε για το λεγόμενο free sharing, για κάτι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να πληρώσει κάποιος, τότε είναι σαν να πληρώνει κανείς. Δηλαδή κάποιος λαμβάνει κάτι δωρεάν γιατί διαθέτει το σώμα του. Αυτό αντιβαίνει στην αρχή που έχουμε ορίσει. Οπότε πρέπει να δούμε κάπως τη διατύπωση. Δεν θέμε να εμποδίσουμε τα ζευγάρια να συνεργαστούν, αλλά όταν πληρώνει κάποιος για το ανθρώπινο σώμα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ε, οι συζητήσεις με την εισηγήτρια νομίζω μας πήγαν προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέτερ Λίζε. Βιτόριο πρώτη κατόπιν. Ε, grazie Presidente. Ε, Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Γιάννα Κουδάκη για την θαυμάσια δουλειά που έκανε και για την, το ανοιχτό της μυαλό κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ποτέ δεν θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από την αρχή της δωρεάν διάθεσης. Ε, θα πρέπει να γίνεται δωρεά τέτοιων ιστών και κιτάρων. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Γιατί αλλιώς ε, θα υπάρξει εμπορευματοποίηση εδώ. Και εδώ οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ σοβαρές. Παραμένει βέβαια το πρόβλημα της συνένεσης στη δωρεά οργάνων. Υπάρχει πρόβλημα για το κατά πόσο είναι δια, διατίθεται αυτό το όργανο εάν το άτομο το οποίο προέρχεται το όργανο δεν έχει εκφράσει τη θέλησή του. μπορούμε να σκεφτούμε ότι η σιωπή είναι συνένεση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε κανονικά πιο σίγουροι από αυτό. Η μια σιγουριά είναι ο θάνατος αυτού του δωρητή. Παραμένει, όπως είπε και ο κύριος Λίζε, του, αυτού του όρου in kind, σε είδος η εισηγήτρια μας εξήγησε ότι πρόκειται για ανταλλαγή οργάνων. Νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτή την ε, ερμηνεία. Αλλά φοβάμαι, φοβάμαι ότι με αυτόν τον τρόπο περνάμε από την πίσω πόρτα, ανοίγουμε μάλλον την πίσω πόρτα στο εμπόριο οργάνων. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτόν τον όρο in kind. Ας προσπαθήσουμε να τον αποφύγουμε, γι' αυτό ακριβώς θα προτείνω μία τροπολογία. Θέλω, έχω ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ομφάλιο λόρο. Έγινε μια τρομερή μάχη δημόσια με διαφημίσεις, ε, μια φοβερή εκστρατεία. Και τώρα αυτή η δωρεά γίνεται ευρέως. Εγώ ήρθα σε επαφή με τους ειδικού και μου είπαν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα του ομφάλιου λόρου. Γιατί? Γιατί τα ομφαλοπλακοντικά κύτταρα ενδέχεται να έχουν βλαστοκύτταρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα από τα βλαστοκύτταρα που μπορούμε να πάρουμε από το ζωντανό άνθρωπο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, πολύ μεγάλη βιβλιογραφία για τα βλαστοκύτταρα από ζωντανού οργανισμού. Αλλά δεν λέει τίποτα βιβλιογραφία ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των βλαστοκυτάρων από τον ομφάλιο λόρο. Από ό,τι ξέρω εγώ λοιπόν, αυτή η μάχη για τον ομφάλιο λόρο εκπορεύεται από την επιθυμία να υπάρξει ένα εμπόριο γύρω από, αυτό το, γύρω από αυτά τα όργανα, ας πούμε. Είναι ενδιαφέροντες οι ομφαλοί λόροι, αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα των βλαστοκυτάρων κατά ανάγκη. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε το θέμα μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί δεν θέλω και με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε πάλι το παραθυράκι στο εμπόριο. Ευχαριστώ, Φρεντερίκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρίνα, την εισηγήτριά μας, για αυτή την έκθεση που Βλέπουμε ήδη ότι δεν είναι τόσο συνενετική ε, όσο φαινόταν στην αρχή. Υπάρχουν έννοιες τις οποίες έχουμε συζητήσει και τις οποίες έχουμε ψηφίσει. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα προβληματικά. Το θέμα αυτής της δωρεάν προσφοράς, ε, της ανωνυμίας. Υπάρχει και το θέμα των, του ιατρικού προσωπικού Τα λόγια εδώ μετράνε. Προσοχή τι γίνεται με την αποζημίωση. Προσοχή με τα λόγια εδώ. Αποζημίωση του δωρητή. Δεν πρόκειται για πληρωμή του δωρητή. Όταν είμαστε δωρητές ε, ιστών ή κιτάρων που, μας, ε, που, που μπορεί να μας ενοχλήσουν πάρα πολύ ως προς την υγεία μας, μπορεί να δικαιούμαστε μια κάποια αποζημίωση. Ε, δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές με αυτό το θέμα. Ε, αυτό που είπε η Μαρίνα για το egg sharing, για την δωρεά ο αρίων. Τι είναι ουσιαστικά ανταλλαγή αρίων είναι. Δεν κατάλαβα. Ας κάνουμε μια πιο ανοιχτή κουβέντα. Τι, ανταλλάσσουμε ένα γαμέτι, μου δεις τον δικό σου, δίνω το δικό μου. Ε, και μάλιστα κάνουμε αυτή την ανταλλαγή, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να πληρώσουμε την θεραπεία. Γλιτώνουμε και τα λεφτά αυτά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για αυτό το θέμα. Για αυτό το σημείο, λοιπόν, 4 και 5, ανησυχώ λιγάκι όλη η αιτιολογική έκθεση που αναφέρεται σε αυτό το σημείο επίση που είναι πολύ περιοριστική, με, με, με ενοχλεί. έχετε πολύ περιοριστική προσέγγιση για την ανταλλαγή γαμετών. Ε, δεν σέβεστε αυτό που συμβαίνει σε 14 κράτη-μέλη, που έχουν πιο ανθρωπιστική, πιο προοδευτική νομοθεσία. Ε, θέλω να, το, τροποποιηθούν αυτά τα σημεία, το λέω ξεκάθαρα, ούτω ώστε όχι να έχω την, να επικρατήσει δική μου φιλοσοφία, αλλά για να υπάρξει μία ισορροπία. Ε, δεν θέλω με το πρόσχημα κάποιου κακώς εννοούμενου ουμανισμού να απορρίψουμε, ας πούμε, ε, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανθρώπους που είναι σε αναμονή κτλ. Και να τους ε, διώξουμε μακριά από τα σύνορά μας. Ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι γίνεται αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει ιατρικός τουρισμός, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. και ξέρουμε ότι μερικές φορές η ανωνυμία είναι ένας τείχος Έχουμε διαφορές λοιπόν σε αυτό το σημείο με την εισηγήτρια. Επίσης, η Μαρίνα είπε στην αρχή ότι η, προ... η προτεραιότητα είναι η δωρεάν προσφορά. Όχι, για μένα το βασικό είναι η ισορροπία. Να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα αυτές τις αρχές και στην έλλειψη αυτών των οργάνων. Δραματική έλλειψη για τους ε, έχοντες ανάγκη, για τους ε, ασθενείς ε, στην Ευρώπη και κυρίως για το μυαλό των οστών, που δεν τον άκουσα πουθενά. Και επίσης ε, πρόβλημα και δραματική έλλειψη γαμετών. Πρέπει να δώσουμε απάντηση σε αυτό το φοβερό ε, ε, πρόβλημα, την έλλειψη αυτή των ιστών και των κιτάρων. Φυσικά, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε καλύτερα τα, τους ανθρώπους ε, ήδη από το 2004 με την πρώτη οδηγία κάναμε μια προσπάθεια να δούμε καταρχάς που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Ε, η, η Κομισιόν μιλάει για την, τον κερατοειδή χιτώνα, μιλάει για το, τους ιστούς δέρματος, μιλάει για τέτοιους ιστούς που μας λείπουν πιο πολύ από άλλους. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, εξυγχρονίσουμε την, το κείμενο του 2004, ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις από τότε μέχρι σήμερα. Εν συνεχεία, αυτά που είπε ο κύριος Πρόντι, που είναι επίσης ουσιαστικά, μπορούμε να ζητήσουμε την Κομισιόν να δεσμευτεί πραγματικά, και το κάναμε μέσω ένα ψήφισμα με τον Πίτερ Λίζε το 2011, για το θέμα του ομφαλοπλακονδιακού αίματος. Δεν είμαι γιατρός. Και γι' αυτό δεν είμαι εμπειρογνώμονα, δεν είμαι επιστήμον. Αλλά είχα μια άλλη ζωή και σε αυτή τη ζωή το επάγγελμά μου ήταν να ακούω αυτού του ανθρώπου του επιστήμονες. Ε, ο κύριος Πρόντιγκ λέει ότι σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει ελπίδα. Όχι, έχω κάνει πάρα πολλές ε, συνεντεύξει με πιονέρους αυτού του θέματο που μου λένε ακριβώ το αντίθετο. Ε, ένα αγόρι, πούμε, στο Βέλγιο, ε, θεραπεύτηκε από μία αρρώστια που δεν ήταν καρκίνος, με τη χρήση αυτών των ε, κυτάρων του ομφαλοπλακουτικού αίματος. Μη λειτουργούμε μόνο με απαγορεύσεις, με περιορισμούς, αλλά με ανθρωπισμό με νομοθεσία, για να πλαισιώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, για να είμαστε προοδευτικοί. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 1% ε, τέτοιου αίματο ομφαλοπλακοντικού συλλέγεται. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά τι δυνατότητε θα είχαμε περισσότερο. Ε, θα ήθελα να επικεντρωθείτε σε αυτό το θέμα στην εκθέσή σα, κυρία Συγγήτρια, γιατί μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Βεβαίω να ευχαριστήσω και την κυρία Γιάννα Κουδάκη για την έκθεση αυτή και για το ότι αντιμετώπισε το θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει όλους τόσο πολύ και από τη συζήτηση αυτή ακούμε πως η συζήτηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί ακόμη και παρά την ε, ευρεία συνένεση. Λέμε όλοι πως πρέπει να δράσουμε ουμανιστικά. Εντάξει, ε, δεν έχει μονοπόλιο κανείς σε αυτό, αλλά το θέμα είναι πως ορίζουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Πρέπει να πάμε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες ε, για να βοηθήσουμε. Υπάρχουν κάποια ηθικά όρια και δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε το τι μπορεί να κάνει κανείς. Υπάρχει νομοθεσία στη Δανία σύμφωνα με την οποία μπορεί κανείς ε, να βοηθήσουν όταν είναι δύο παιδιά, δύο αδέρφια, το ένα να βοηθήσει το άλλο με κάποια ε, δωρεά. Αλλά ε, εντάξει, υπάρχει, το, υπάρχει περίπτωση του να, να γεννηθεί ένα παιδί για αυτό τον ε, σκοπό. Ε, τι είναι, το δεύτερο παιδί είναι ανταλλακτικό του πρώτου. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τα, τα όρια μας. Οπότε πρέπει να είναι, όπως είπαμε, εθελοντική και δωρεάν η προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Παρόλα αυτά βεβαίως ε, υπάρχουν ε, διάφορες ε, περιπτώσεις. Υπάρχει πάλι και το παράδειγμα του 2007 στη Δανία. Σε όλα τα ΜΜΕ εμφανίστηκε μία γυναίκα άνω των 60 που έμεινε έγκυος βεβαίως με τέτοια μέσα. Και συζήτησαν μετά στη Δανία και λέγανε «Ε, μεγάλοι άντρες σε αυτή την ηλικία έχουν παιδιά. Γιατί να μην κάνουν και οι γυναίκες σε αυτή την ηλικία παιδιά. Ε, Βεβαίω, εντάξει, καλό είναι να μην έχουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία παιδιά, θέμε και το όφελο των παιδιών, να έχουν υγιείς, ε, γονεί. Ε, γονείς. Αλλά αυτά τα πράγματα Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν ήταν φυσική διαδικασία. Πήγε στην Αγγλία και βρήκε αγγλικό άριο. Εγώ ρώτησα την Κομισιόν, η Κομισιόν ρώτησε στην Αγγλία και τους λένε αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Εμφυτεύουμε οάρια και σε γυρές κυρίες. Τίποτα παραπάνω δεν ξέρουμε. Αλλά ε, οπωσδήποτε κάπως έγινε αυτή η υπόθεση και κάπως το βρήκε αυτό το Άριο. Ποια γυναίκα θα έδινε ο Άριο εθελοντικά εάν ήξερε πως ε, θα πήγαινε σε μια γιαγιά εάν θέλετε η οποία ήθελε να γίνει μητέρα. Οπότε ε, Βλέπετε, δεν πρέπει να υπάρχουν ανταλλάγματα και μετά τι είπαν από την Αγγλία δεν, ήταν, δεν υπήρχε αντάλλαγμα τελικά όμως είχε πληρωθεί η άλλη γυναίκα οπότε πρέπει να ε, διατηρήσουμε μια ανθρωπιστική ε, στάση και να φροντίσουμε να είναι όλα αυτά τα πράγματα εθελοντικά όπως είπα και χωρίς ανταμοιβή. Για την αμοιβαιότητα τώρα που λέγατε, την ανταλλαγή, και αυτό προβληματικό είναι. Αν μια γυναίκα θέλει να δωρήσει ένα οάριο και μας δίνετε εσείς το σπέρμα σας, Τι, εντάξει, αν μια γυναίκα, ξέρω εγώ, δεν είναι αρκετά γόνιμη, ε, μπορεί να απευθυνθεί στην, ε, στην αδερφή της, να γίνεται εντός της οικογένειας. Δεν λέω να μην υπάρχουν δωρεές, αλλά ε, δεν μπορούμε βεβαίω και να πάρουμε το αυγό κάποιου, κάποιας, το, το, το άριο κάποιος με συγχωρείτε, χωρίς τη, τη θέλησή της. και ε, όσον αφορά τώρα τις θεραπείες αυτές γονιμότητας που δεν θα τις αποφύγουμε και αυτές πρέπει να μπορούμε και στην ε, Επιτροπή μας ε, να δούμε το ζήτημα της υπογονιμότητας των ανδρών. Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχει αυξηθεί πολύ η υπογονιμότητα ανδρών και γυναικών. Και πρέπει να δούμε την αιτία. Όχι μόνο το σύμπτωμα να θεραπεύουμε. Μετά, έχουμε το ζήτημα του αίματος από τον ομφάλιο λόρο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μας υπόσχονται διάφορα ότι θα είναι θαυματουργό και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Δεν ξέρουμε εάν μια θεραπεία θα μπορέσει ποτέ να αναπτυχθεί από τα βλαστοκύτταρα του αίματος αυτού. Εντάξει, μην ε, επενδύσουμε και όλες μας ελπίδες εκεί πέρα και υποσχεθούμε στους γονείς πως θα θεραπεύουν το γονείς τους στο μέλλον ότι θα έχει κάπου ανταλλακτικά δηλαδή το παιδί γιατί πληρώνουν πάρα πολλά για να αποθηκεύσουν αυτό το αίμα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. είναι πάρα πολύ χρήσιμο βεβαίω να υπάρχουν αυτές οι τράπεζες και όσο πιο ευρωπαϊκά τόσο το καλύτερο. Να ανταλλάσσουμε και μεταξύ μας τους πόρους, να υπάρξει μια δικτύωση. Αλλά στη Δανία σημαίνει το εξής. Αυτό γίνεται μέσω μιας δημόσιας διοίκησης και όχι μέσω του ιδιωτικού τομέα για να υπάρξει μια ισότιμη αντιμετώπιση των ασθενών ε, και να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Τρεις ομιλητές έχουμε τώρα στον κατάλογο και μετά θα κλείσει ο κατάλογος. Γκροστέτ, Λίντα Μακάβαν και Ντάγμαρ Ροτ Μπέρεντ τρία λεπτάκια περίπου η κάθε μία για να έχουμε χρόνο να πει και η Κομισιόν ε, κάτι και να απαντήσει στην εισηγητρία. Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να, ειση... να συγχαρώ την κυρία Γιανακουδάκη για την ποιοτική της έκθεση. Ποτέ δεν έχουμε πολύ χρόνο αλλά θέλω να μιλήσω για ένα πρόβλημα που με απασχολεί εδώ και χρόνια. Πρόκειται για τα κύτταρα του ομφάλιου λόρου και τα κύτταρα του ομφαλοπλακοντιακού αίματος. Δεν συμφωνώ με τους απρόθυμους συναδέλφους μου. Βρίσκω πολύ σοβαρό και απαράδεκτο σήμερα που θεωρούμε ότι ο ομφάλιος λόρος είναι κάτι που πρέπει να πεταχτεί στον κάδο του νοσοκομείου. Ενώ είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να βρούμε νέες θεραπείες, είμαι πεπισμένη ότι σε λίγα χρόνια, πόσα χρόνια τώρα θα δούμε, μπορεί να είναι και μερικές δεκαετίες, δεν θα έχουμε ένα φάρμακο για όλο τον πληθυσμό, αλλά θα έχουμε φάρμακα ή θεραπείες εξατομικευμένες και που θα μας επιτρέπουν να θεραπεύσουμε ασθένειες που σήμερα δεν είμαστε σε θέση να θεραπεύσουμε. Παρότι η έρευνα εξελίσσεται πολύ, σε αυτόν τον τομέα εξελίσσεται αλματοδός. Παρότι δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα που έχουμε. Και λυπάμαι που σε μια χώρα όπως η δική μου, που έχει νοσοκομεία, πολύ άριθμα, μη τι άλλο, συστηματικά να πετάμε όχι μόνο το φαλοπλακοντιακό αίμα, αλλά και τον ίδιο τον λόρο. Γιατί ξέρουμε ότι κάποια κύτταρα βρίσκονται στον ομφάλιο λόρο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για να προχωρήσουμε με αυτές τις θεραπείες. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ε, απόβλητο ο ομφάλιος λόρος. Θα πρέπει να το βάζουμε σε τράπεζες. Ε, ξέρουμε ότι έχουμε μια προθεσμία 24 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου για να μεταφέρουμε τον ομφάλιο λόρο και το αίμα του ομφάλιου λόρου. Ε, μέσα σε 24 ώρες με τα αεροπλάνα πάμε γρήγορα και πολύ μακριά και μπορούμε να στείλουμε τον ομφάλιο λόρο σε τράπεζες. Δημόσιες τράπεζες φυσικά. Τώρα, αν δεχτούμε και τι ιδιωτικέ, θα πρέπει οι κανόνε και οι προποθέσει να είναι πολύ αυστηρέ, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια ιατρική δύο ταχυτήτων. Μία για του πλούσιου που θα έχουν ιδιωτικέ τράπεζε και οι υπόλοιποι δεν θα έχουν τίποτα. Θέλω λοιπόν να τονίσω αυτό το θέμα, γιατί χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρόνια, χάνουμε προοπτικές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν πριν από λίγο καιρό τη έθεσα το ερώτημα. Θα πρέπει, τη ζήτησα μάλλον να ετοιμάσει μία ανακοίνωση, ούτω ώστε όλα τα κράτη-μέλη να ανακτούν και να αποθηκεύουν το αίμα των φάλιου λόρου και τον ίδιο τον ομφάλιο λόρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίντα Μακάβα και μετά. Και μετά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Και ευχαριστώ για ερώτηση. Θέλω να πω κάτι για το οποίο, το οποίο έδειξε ο Πίτερ Λίζε αυτό το θέμα της εθελούσιας δωρεάς των ε, οαρίων όσον αφορά την αγωγή in πριν από λίγα χρόνια πριν εσύ η συγκήτρια είχαμε κάποιες κυρίες οι οποίες και καλύπτονται από αυτή την αμοιβή σε είδος σε κάποια κλινική, σε κάποια τράπεζα και όταν είδαμε τι αξίζουν αυτές οι δωρεές ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Δηλαδή, η δωρεά των αρίων δεν είναι κάτι το ασήμαντο. Πρόκειται για μία επέμβαση μίζωνος σημασίας με κίνδυνο υγείας. Είναι πράξη αλτρουιστική. Γιατί κάποια γυναίκα 22 ετών στη Ρουμανία πούμε, να, κάνει έτσι μια δωρεά. Μα είναι πολύ σπουδαίο. Το είπαμε και το ξαναείπαμε, έγινε τελικά μια ευρύτατη συζήτηση. Είπαμε, μίλησαμε για τη γονιμότητα και έτσι ε, έχουμε επομένως διαφορετικούς διάβλους που φτάνουν αυτά στην Ευρώπη και άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα συζητούμε όλα αυτά και προσοχή να μην ανοίγουμε κερκόπορτες ούτως ώστε κάποιοι νέοι άνθρωποι να υφίστανται εκμετάλλευση. Γιατί σας είπα, δεν είναι ασήμαντη υπόθεση αυτή. Μπορεί να θέσει εν κινδύνο μακροπρόθεσμα την υγεία κάποιου. Άρα, μεγάλη προσοχή στο πώς διατυπώνουμε τέτοια νομοθετήματα. Ευχαριστούμε, Λίντα. Ντάγμαρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ξέρουμε εδώ και χρόνια πως το ζήτημα της ε, δωρεάς οργάνων ε, και ιστών και κιτάρων είναι ευαίσθητο. Ο Φεντερίκ είπε πως πρέπει να ξαναδούμε την παλιά νομοθεσία ίσως. Ε, εγώ θέλω να σας αποτρέψω, ήμουν τότε η εισηγήτρια και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η νομοθεσία. Ρωτήστε και τον κύριο Νικολασίτς. Δεν συζητήσαμε τέτοια ζητήματα. Μιλούσαμε μόνο για βλαστοκύτταρα των ε, εμβρίων και η συζήτηση ήταν ε, θα δημιουργήσουμε τέρατα. Αυτό λέγαμε τότε μόνο. Είχαμε λοιπόν εύρωστη νομοθεσία και το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη και το τι θέλουμε. Τι γίνεται στα κράτη. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, απλούστατα, από το ένα στο άλλο. Ε, όταν συζητάμε αυτό το θέμα, πρέπει να έχουμε κάποτε και το θάρρος εμείς να κάνουμε μια ηθική αξιολόγηση. Παραδείγματος χάρη, δωρεά ενός οαρίου που συνδέεται με μεγάλους κινδύνους, με ορμόνες και τέτοια, είναι καλύτερο ή χειρότερο από το να δώσει κανείς νοτιέο ε, νοτιαίο όχι μυαλό των οστών, ε, των οστών, για να καταπολεμηθεί ο καρκίνος του αίματος. Αξίζει περισσότερο ή λιγότερο. Θα αποφασίσουμε εμείς και θα πούμε πως ε, κάποιος ο οποίος βοηθάει έναν άνθρωπο με καρκίνο αξίζει και κάποιος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να, σε κάποιον άλλο να μπει έγκυος αξίζει λιγότερο και τα δύο ε, είναι ζητήματα για την υγεία δεν το συζητάμε και μετά αφηρούμε εντάξει τώρα δεν, δεν το συζητάμε για προσφορά αίματος και σπέρματος αυτά είναι αυτονόητα όταν ακούω λοιπόν τους συναδέλφους Ε, οι γονεί που έχουν ένα στο παιδί υποφέρουν, υποφέρουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει νόμος που θα επιτρέψει σε γονείς να κάνουν ανταλλακτικό παιδί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα, στην Κίνα ίσως. Δεν λέει κάποιος ε, επιτρέπεται ή όχι να κάνετε ένα άλλο παιδί ή όχι. Το θέμα είναι αν επιτρέπεται από ένα ανήλικο παιδί να αφαιρέσουμε ιστό. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτή τη θέση αυτών των γονιών που πρέπει να λάβουν αυτή την απόφαση. Να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα νεφρό, ένα νεφρό, κάτι τέτοιο για, να σώσουν το άλλο παιδί. Κανείς στον κόσμο δεν δε, θέλει να λάβει τέτοια απόφαση. Οπότε ο τόνος με τον οποίο το συζητάμε ε, με, με, με, με πληγώνει. Αυτό το οποίο θεωρώ πως πρέπει να τονίσουμε είναι το ζήτημα τι ευκαιρίες προσφέρουμε στους δωρητές ε, κιτάρων και ιστών. Και επειδή Φρανσουάζ ανέφερε το αίμα του ομφάλιου λόρου, έχει δίκιο. Θα έχουμε σε λίγο προσωπικά φάρμακα. Φάρμακα τα οποία... Ναι, ναι, θα σταματήσω. Φάρμακα για λίγους ανθρώπους. Ε, εννοώ κομμένα στα μέτρα τους. Και αυτό είναι καλό. Τώρα, εγώ δεν θέλω να έχω ιδιωτικέ τέτοιε τράπεζε. Δεν θέλω να γίνει βιομηχανία. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, να τα βάζουν ε, κάποιοι άνθρωποι στην άκρη ε, αν είναι δηλαδή, αν υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον να έχουν καλύτερη θεραπεία, έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλους. Ε, εγώ αυτό θα ήθελα να, να δω. Ευχαριστώ. Dagmar roth ε, Να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν για πέντε λεπτά και ξέρω πως είναι δύσκολο, είναι σημαντική η συζήτηση. Ε, καλή νομίζω συζήτηση αυτή που είχα. Τώρα να ακούσουμε την Κομισιόν και μετά την εισηγητρία. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε τη δουλειά της εισηγήτριας. Έκανε πολλή προσπάθεια, εξόδεψε χρόνο και αν δείτε το αποτέλεσμα συνειδητοποιείτε ότι είναι καλή η ισορροπία της έκθεσης δεδομένης της περιπλοκότητας των θεμάτων, όπως φάνηκε τη συζήτηση. συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου πλευράς Κομισιόν, ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της προσφοράς νέων και καλών θεραπείων στους πολίτες και από την άλλη αυτό να μην έχει ως κόστος την εκμετάλλευση του ανθρώπινου σώματος, την εμπορευματοποίηση και ενδεχομένως το λαθρεμπόριο. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στην ασφάλεια και στην ποιότητα και πολλές από τις αρχές που συζητάμε μέχρι στιγμής εμπίπτουν δυστυχώς στις αρμοδιότητες των κρατών μελών ε, το οποίο περιπλέκει περαιτέρω τη συζήτηση ειδικά όταν μιλάμε για αποζημίωση και τη σχέση ανάμεσα στην αποζημίωση και στην πληρωμή σε διαφορετικά κρατημέλη οι συζητήσεις αυτές παίρνουν διαφορετικούς δρόμους. Χαιρόμαστε που η έκθεση εστιάζεται σε κάποια βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά, την χρησιμότητα, την διαφάνεια, που μπορεί να διασκεδάσει πολλές από τις ανησυχίες που έχουμε. Χαιρόμαστε επίσης που το θέμα του ομφαλοπλακοντιακού αίματος ε, τέθηκε ρητά. Και κάποιες από τις προτάσεις που κάνετε σχετικά είναι πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικό για τον ομφάλιο λόρο και τα βλαστοκύτταρα να ξεχνάμε, να θυμόμαστε μάλλον, ότι δεν πρόκειται για εμβριακά κύτταρα, γιατί μερικές φορές περιπλέκεται η συζήτηση ε, λόγω αυτού του θέματος. Δεν μιλάμε για αυτά τα κύτταρα, μιλάμε για τα, για τα ε, κύτταρα του αίματος που θεραπεύουν λευχαιμία ή τεσμο, βοηθάνε με τις θεραπείες ε, καρκίνου και λευχαιμίας και μπορεί να δημιουργήσουν και νέες θεραπείες. Αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Το δυναμικό είναι δυναμικό, δεν είναι πραγματικότητα. Θα πρέπει να ενημερώνετε το κοινό. Το σημείο 16 για την ε, αφύπνιση και την ενημέρωση και τις εξαρτίες πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικό. Το εμφαλοπλακοντιακό αίμα δεν έχει να κάνει με το κατά πόσον θα έχουμε εθνικ... δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, αυτό είναι εθνική απόφαση. Αλλά ότι χρειαζόμαστε ένα καλό πλαίσιο για την ασφάλεια και την ποιότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα βλαστοκύτταρα, είτε έχουμε να κάνουμε με ιδιωτικούς είτε με δημόσιους φορείς. Η Κομισιόν σκέφτεται κάποια project για να προωθήσει αυτό το θέμα θα πρέπει λοιπόν όλοι οι φορείς να έχουν και να σέβονται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Ο στόχος με το εμφαλοπλακονδιακό αίμα επίσης είναι να υπάρχει δημόσια, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες στους πολίτες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι το απόσταγμα της έκθεσης και νομίζω ότι στο σημείο 18 το απεικονίζει πολύ ωραία η συγγήτρια. Περιμένουμε λοιπόν την τελική έκθεση που θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο και Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε την Επιτροπή των Κρατών Μελών, όπου συμμετέχουν οι εμπειρογνώμες των κρατών μελών. Θα ήθελα όταν ολοκληρώσει και αποκρισταλώσει την έκθεσή της η συγγήτρια να έρθει εκεί με την έκθεση αυτή στην Επιτροπή, για να το συζητήσουν οι εμπειρογνώμε των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω γρήγορα. Τα εύκολα πρώτα. Ε, η αποζημίωση σε είδο. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για χρήματα, για ανταλλαγή οργάνων. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε. Και οποιαδήποτε τροπολογία το διευκρινίζει είναι καλή. Ε, και θα το βγάλω αν δεν διευκρινίζεται παρκώ. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι γαμέτης για γαμέτη και ότι βοηθούν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Εθελοντική δωρεά. Ναι, είναι εθελοντική, αλλά φυσικά ε, το κόστος καλύπτεται για ιατρικά έξοδα, για απώλεια εισοδήματο, για ταξιδιωτικά έξοδα κτλ. Δεν θέλω δηλαδή να περιορίσουμε του ανθρώπου να κάνουν δωρεές, ε, θέλω να τους βοηθήσω. Ε, ορισμένοι αναφέραν ε, τη σημασία επίσης του μυελού των οστών για τα βλαστοκύτταρα. Εμεί έχουμε ένα ίδρυμα ε, όπου κατατίθεται τέτοιο, τέτοιος μυελός των οροστών, γιατί τα βλεφτοκέντρα είναι πολύ σημαντικά. Έπειτα, ε, για το νεφρό, δύσκολο ιστός, δύσκολο είναι να ξεφύγουμε από τα λεφτά. Επίσης, ε, τα οάρια. Ε, τα οάρια γίνονται μωρά. Είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες. Πρέπει να δούμε τι, θα, τι, μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα. Τα πιο προβληματικά ε, είναι το ομφαλοπλακοντιακό αίμα. Ε, εγώ μίλησα με ειδικού στη Ρώμα τον κύριο Νάνο ή Νάνη, ένα συμπαθητικό άνθρωπο, ο οποίος ε, στην αρχή ήταν κατά αυτού του αίματο. Αλλά μετά μου είπε ότι αντίθετα ήθελε. Ήταν θέμα ότι δεν υπάρχει αρκετό τέτοιο αίμα, ε, ώστε να, να αξίζει τον κόμμα, το έχουν όλοι. Θα πρέπει να δούμε ε, αυτό που υπάρχει, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει επίσης ε, Είναι σημαντικό να υπάρχουν και ιδιωτικοί φορεί ε, συλλογή τέτοιου αίματος. Αυτό σε σημαντικέ. Μην ξεχνάτε ότι δημόσια ε, τέτοιοι φορεί γίνεται μόνο στις μεγάλες πόλεις. Ε, ξέρω ότι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έχω Αλλά θέλουμε και ιδιωτικού φορεί που συλλέγουν γρήγορα αυτό το αίμα και βοηθούν την, τα εθνικά συστήματα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και θα πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά υποστηρικτικά, όχι για τα λεφτά. Ξέρω ότι γίνεται μια συζήτηση για το πόσο σημαντικό είναι το αίμα αυτό. Ε, είναι χρήσιμο για τα αδέρφια, είναι χρήσιμο για το παιδί. Ε, δεν έχει αποφασιστεί αυτό, συζητιέται. Ε, δεν θέλω να κλείσω καμία πόρτα όμως, ε, αν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουμε ένα παιδί. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα ανεξερεύνητα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο στην Επιτροπή. Ε, ίσως πρέπει να μετακινήσουμε την ημερομηνία, να έχουμε περισσότερο χρόνο θα πρέπει, όπως είπε και η Ντάγμαρ, να τα δούμε αυτά ως ευκαιρίες. Ευκαιρία σημαίνει καλύτερο σύστημα, βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και είναι άρρωστοι. Περιμένω τις τροπολογίε για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ, κυρία Γιανακουδάκη. Νομίζω πως είχαμε μια καλή συζήτηση. Αναδείξαμε όλες τις πτυχές του θέματος προθεσμία για τροπολογίες είναι η 3 Μαΐου ζητήσατε αναβολή της προθεσμίας αυτό σημαίνει πως το χρονοδιαγραμμά μας θα πάει όλο το χρονοδιάγραμμα πίσω το πατήσετε το μικρόφωνο Μήπω μπορείτε να μα δώσετε μια εβδομάδα παραπάνω για τι τροπολογίε γιατί είναι πράσινη εβδομάδα την επόμενη, επόμενη εβδομάδα και έχουμε ψηφοφορία τον Ιούνιο. Εάν θέλετε αναβολή μια εβδομάδα, τότε αυτοδικαίω πάμε για ψήφιση τον Ιούνιο. Εντάξει, εντάξει, λέει κύριε Γεννατάκη. Συμφωνούν οι σκιώδε συζητητέ. Εάν όλοι οι σκιώδε συζητητέ συμφωνούν, τότε αυτό θα κάνουμε. Θα ψηφίσουμε τον αναβάλλεται και πάμε το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Πάμε παρακαλώ. Το επόμενο σημείο είναι το υπαριθμό 21. Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η εισηγήτρια είναι η συνάδελφος Γκαρδίνη. Έχετε εσείς τον λόγο να μας κάνετε μια εισαγωγή. Κυρία Ευχαριστώ. η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για μια ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν και ξεκινήσαμε την δουλειά ήδη, κάναμε διάφορες συναντήσεις, όπου ε, συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι Θα είμαι πολύ σύντομη σε αυτή την παρουσίαση, γιατί το πιο ενδιαφέρον θέμα είναι το να μπορέσω εγώ να ακούσω τη θέση των διαφόρων ομάδων, των διαφόρων πολιτικών οικογενειών και των διαφόρων χωρών στο, που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο, το κοινό μας σπίτι. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι όταν ψηφίσαμε το Σεπτέμβρη την ε, έκθεση για να δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Καταστροφές, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Καταστροφές, είχαμε μια συντριπτική πλειοψηφία. Ε, το κείμενο αυτό καλύπτει τα αιτήματα του 90% των Ευρωπαίων πολιτών, όπως μας τα διατύπωναν μέσα από το Ευρωβαρόμετρο, που θέλουν περισσότερα από την Ευρώπη. Πολίτες που θέλουν περισσότερα από την Ευρώπη, ε, για την αντιμετώπιση των καταστροφών, όλων των καταστροφών, ή οδήποτε είδους. Μεγάλες καταστροφές που λόγω επικουρικότητας δεν μπορούν να τις διαχειριστούμε σε περιφερειακό επίπεδο. Η Κομισιόν λοιπόν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας και βγήκε η πρότασή της στο στα τέλη του 2011. Είχαμε λοιπόν όλο το χρόνο να μελετήσουμε πολύ αναλυτικά την πρόταση της Κομισιόν Ανασημείου. Φυσικά, όπως πάντα, είναι βελτιώσιμη. Για ορισμένα σημεία πρέπει να τα τροποποιήσουμε, να τα εμβαθύνουμε, να τα διευκρινίσουμε. Γιατί γίνουν κάποιες ανησυχίες ορισμένα σημεία, όντως, σε κάποια κράτη-μέλη. Ανάλογα με την δομή του κάθε κράτους. Αλλά με σεβασμό των δομών του κάθε κράτους μπορούμε να διορθώσουμε το κείμενο, να το προσαρμόσουμε, ούτως ώστε να καλύπτει και τις 27 διαφορετικές χώρες. Μην ε, ξεχνάτε ότι και ο όρος ε, πολιτική προστασία δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην Ιταλία, στη χώρα μου, ακόμα και στο δημοτικό και στον υπηαγωγείο μιλάμε για πολιτική προστασία. Αλλά υπάρχουν χώρες όπου αυτός ο όρος, παρότι μιλάει για βοήθεια, δεν ονομάζεται έτσι παντού υπάρχει προβλέπεται η βοήθεια ας πούμε, των πολιτών σε περίπτωση καταστροφών, αλλά δεν χρησιμοποιείται ο όρος αυτός, πολιτική προστασία. Ε, το βασικό είναι να περάσει όμως ένα κοινό όραμα ευρωπαϊκό. Είδαμε λοιπόν κάποια βλέμματα λίγο ανήσυχα να εμφανίζονται από εδώ και από εκεί. Όχι με επίσημο τρόπο, αλλά όλα εξαρτώνται από αυτό νομίζω. Μην ξεχνάμε την σχεδόν ομόφωνη ψήφο του περασμένου Σεπτέμβρη με δεδομένο αυτό νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε επί του περιεχομένου. Συμφωνούμε όλοι με τον στόχο. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι μια θαυμάσια βάση για να δουλέψουμε, για να προχωρήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ε, μην ξεχνάτε, υπενθυμίζω, ότι ο πυρήνας της είναι να περάσουμε από μια απάντηση ad hoc ανακαταστροφή σε ένα σύστημα όπου προληπτικά έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα μέσα όλα τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να προγραμματίσουν τις ε, πιθανές τους παρεμβάσεις. Να υπενθυμίσω ότι η πολιτική προστασία ήταν και θα παραμείνει εθνική αρμοδιότητα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε αυτό το γεγονός. Έχουμε στεναρές βάσεις νομικές όμως. Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας Η πολιτική προστασία λοιπόν υπάρχει, υπάρχει και νομική βάση και το κείμενο αυτό είναι το απόσταγμα ετών εμπειρίας στον τομέα αυτό. Ένα θαυμάσιο κείμενο εργασίας. Το θέμα της πρόληψης είναι καινούριο κεφάλαιο και της προετοιμασίας. Πρέπει να τα ενισχύσουμε θα υπάρξει αυτό το νέο κέντρο ανταπόκρισης σε κατεπίγουσε ανάγκες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χρειάζεται για να γίνουν όλα πολύ πιο γρήγορα, αποτελεσματικά, λιγότερο γραφειοκρατικά. Υπάρχουν και άλλα ευαίσθητα σημεία που αφορούν τη χρηματοδότηση βέβαια. Τη διαχείριση του κινδύνου την δημιουργία αυτών των ομάδων, αυτών των πουλ, των ομάδων αυτών έτοιμων στα κράτη-μέλη που μπορούν να κινητοποιηθούν ανα πάσα στιγμή. Υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορούμε να εμβαθύνουμε βέβαια. Αλλά μην χάσουμε την ευκαιρία με αυτό το εργαλείο να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες το όραμα μιας Ευρώπης που είναι στο πλευρό τους. Μια Ευρώπη που είναι μέσα στην καθημερινότητά τους. Μέσα από όλες αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης, μέσα από όλα αυτά τα φυλάδια που κυκλοφορούν από τον υπηαγωγείο σχεδόν και το... και με αυτό το νούμερο 112 ε, αυτή την ειδική γραμμή, ας πούμε την τηλεφωνική που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, θέλουμε να τους δώσουμε αυτή την ιδέα της ε, Ευρώπης που είναι κοντινή σε αυτού. Ελπίζω να συνεχίσουμε την πολύ επικοδομητική συνεργασία με την Κομισιόν, όπως κάναμε και το 2011. Ευχαριστώ. Η πρώτα ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Πρόεδρε. Και εμείς θεωρούμε θετική την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία πέραν όλων των άλλων μας δείχνει το δρόμο για μια λύση. Μια λύση για πρόβλημα που μας απασχολεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια. δούμε επίση πάρα πολύ θετικό το ότι αυτή η πρόταση απλουστεύει τα υπάρχοντα νομοθετήματα και μέσα πολιτικής. Έτσι αναβαθμίζεται η ευρωπαϊκή συνεργασία. Κατά αυτόν τον τρόπο είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την ε, αντίδρασή μας κάθε φορά που υπάρχει κάποια φυσική καταστροφή, κάποια θεομηνία. Αυτό αφορά επίσης και τα θέματα περικοδότησης, χρηματοδότησης. Και σε αυτό το επίπεδο θεωρούμε ότι όπως έχουμε στο καινούργιο κεφάλαιο κάλυψη όλων αυτών των ε, ζητημάτων νομίζουμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται πιο ολοκληρωμένα. Οπότε έτσι είναι σε θέση τα κρατη να αναβάνουν σχετική πρωτοβουλία, ε, μπορούν να έχουν υποστήριξη οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δραστηριότητες που έχουν σχέση με τέτοια φαινόμενα. Ε, φυσικά πρόκειται περί συγχρηματοδότηση, εμπλέκονται εδώ και τα κρατημέλη, κυρίω στα θέματα τη μεταφοράς. Όσον αφορά τώρα τις ε, δημοσιονομικέ διατάξεις, στα πλαίσια του πολιετούς πλαισίου 14-20, θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Επίσης, θεωρούμε ότι το έγγραφο αυτό είναι συνδεταγμένο και διαρθρωμένο πάρα πολύ ολοκληρωμένα και τα λέει όλα ξεκάθαρα. Έχει τέσσερις άξονες, πρόληψη, εκ των υστέρων επέμβαση, εξωτερική διάσταση, ανταπόκριση και έχουμε βέβαια και τις δημοσιονομικές διατάξεις που είναι σε χωριστό κεφάλαιο. Επομένως, συμπερασματικά εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία πάρα τα οποία βγαίνουν μέσα από αυτή την πρόταση. Επίσης, θεωρούμε ότι παρέχονται εγγυήσεις για έναν καλύτερο συντονισμό, για μια αντίδραση ταχύτερη και πιο αποτελεσματική των κρατών μελών. Και επίσης και εξωτερική διάσταση καλύπτεται όπως πρέπει. υπάρχει κάποια συνέπεια, κάποια συνέργεια των προσπαθειών σε διεθνέ επίπεδο. Έχουμε επίσης κάποια αρρωγή μέσω του σχετικού μηχανισμού και από τα, ε, Ηνωμένα, ή Έθνη. Βεβαίως να βάλετε υπόψη και, και η αρχή της αναλογικότητας αλλά και της επικουρικότητας. Και αυτό κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ επενετό. Όμω πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση. Πρόκειται για μια αξιόλογη αφετηρία για να εργαστούμε και επομένω κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες του θέματος στη συνέχεια και ο καθένας να κατεβάσει τις τροπολογίες του, τις προτάσεις του και τις ιδέες του. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε πρεμιέρα εδώ πέρα. Μια νέα συνάδελφο που χαιρετήσαμε χθες κυρία Τάιλερ, η οποία είναι και σκιώδης εισηγήτρια. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ξόνομα των φιλελευθέρων καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν. Είναι λογικό να διδασκόμαστε από τις εμπειρίες των τελευταίων ετών έτσι που είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι για τι φυσικέ καταστροφέ. Και επίση έχουμε και το θέμα τη πρόληψης που είναι ένα καινούριο κεφάλαιο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Είπαμε επομένω ότι οι προσδοκίε υπάρχουν όσον αφορά μια καλύτερη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχουμε πλημμύρε ή άλλου είδου φυσικέ καταστροφέ στα κράτη-μέλη. Ο κόσμο αυτό προσδοκά. Περιμένει. Ο ένα να βοηθάει τον άλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και εμεί περιμένουμε πώ και πώ το σχέδιο έξω από την κυρία Καρδίνη. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο κατάλογος. Η κυρία Γκροστέτ που είχε ζητήσει το λόγο. Ε, έχετε πολύ χρόνο. Όσο χρόνο θέλετε. Οτιδήποτε δεν είχατε πει αυτή τη βδομάδα, πείτε τα τώρα. Μην ανησυχείτε, σύντομη θα είναι. Ήδη τα συζητήσαμε αυτά στην έκθεση πρωτοβουλίας της ε, Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη το 2011 και είχα υπενθυμίσει τότε ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη ε, δυνατότητα αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνουμε την ε, μετακίνηση των πόρων και των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική προστασία και την πολιτική προστασία. Θυμάμαι την έκθεση Μπαγνιέ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπενθυμίζει διάφορα στοιχεία και είμαι πεπισμένη ότι στην έκθεση του, της συναδέλφου κυρίας Γκαρντίνη θα ξαναβρούμε αυτά τα στοιχεία. Υπενθυμίζω ποια είναι. Καταρχάς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη σπατάλη, για να το πω έτσι, και σε ανθρώπινο επίπεδο και σε επίπεδο οικονομικό. Κάνουμε τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει συντονισμό, δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη βάση από κάτω προς τα πάνω επί τη βάση του εθελοντισμού και ανάλογα με την εξειδίκευση του κάθε κράτου μέλου. Θα πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη μα την ικανότητα αντίδραση που να βασίζεται στις, και στι ικανότητε των υπερπεριφερειακών περιοχών και στι απομα... απομακρυσμένε απομακρυσμένες ε, περιοχές που συνήθω είναι πολύ μακριά από την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όπω είπε η κυρία Γκαρντίνη, όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σεβασμό τη αρχή επικουρικότητα, όχι μόνο τη επικουρικότητα των κρατών μελών, αλλά και του ΟΗΕ. Ούτως ή άλλως έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο εκεί. Γιατί έχουμε αυτό το νούμερο ε, για τα κατεπήγοντα 112. Να, κάτι που κάναμε. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε και την προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες. Και αυτό μέσω της διπλωματικής και προξενικής προστασίας. Είμαι πεπισμένη ότι όλα αυτά τα σημεία θα ενσωματωθούν στην έκθεση Γκαρδίνη. Να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτή η έκθεση Μπαρνιέ είναι μια καλή βάση προβληματισμού για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε την Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που συναποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναλάβω πως η Κομισιόν αναμένει τη συνεργασία μαζί σας και με την Επιτροπή σας. Επίσης, στηρίζουμε πλήρω την Επιτροπή στο στόχο της να έχει ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα στον τομέα αυτών, ένα σημαντικό τομέα για τους πολίτες, όπως είπε η κυρία και για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τα πρόσφατα ευρωμαβαρόμετρα έδειξαν πως οι πολίτες στηρίζουν αυτή την υπόθεση και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε φιλόδοξες συμφωνίες μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και γρήγορα. Να επαναλάβω τα τρία βασικά στοιχεία της πρότασης αυτής ε, κατά την άποψή της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα η πρόταση σέβεται την επικουρικότητα και το σημαντικό ρόλο που παίζουν τοπικές και περιφερειακές αρχές όταν μιλάμε για την προστασία των πολιτών. Αφεντηρία μας είναι πως οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ε, είναι αυτές που αντιδρούν καλύτερα σε μια καταστροφή. Και αυτό βέβαια είναι η βάση της πρότασής μας. Ρόλος της Ένωσης είναι να στηρίζει, να συμπληρώνει και να συντονίζει και αυτούς τους τομείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Κατόπιν για την πρόληψη πρέπει να γίνει ένα βήμα να έχουμε πιο συγκεκριμένους κανόνες για την πρόληψη των καταστροφών οπότε έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση προετοιμασία δηλαδή για τις καταστροφές αλλά και τι μπορεί να γίνει για να τις προλάβουμε τέλος ενισχύουμε την προετοιμασία μέσω των απαραίτητων εργαλείων και μέσων για να μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα. Η πρόταση εθελοντικής ε, συνένωσης των μέσων ε, όπου υπάρχουν κενά είναι ε, σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν μια κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω και βασιζόμαστε στα υφιστάμενα μέσα των κρατών μελών και τις εθελοντικές ε, δεσμεύσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε τον εθελοντικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν πολλές ε, υποχρεώσεις στην νομοθεσία, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να γίνει ένα βήμα παρακάτω μαζί με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε αναμένουμε τη συνεργασία μαζί σας και ελπίζουμε να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό σύντομα. Ευχαριστώ. Καλώς ορίζω για την Προεδρία της Δανίας. Χαίρομαι που είστε εδώ. Και θα τοποθετηθείτε και στο θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη θαυμάσια συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και όπως ε, σας είπατε, είναι η... Ε, σας είπε η Κομισιόν, η πρώτη φορά που συναποφασίζεται για αυτό το νέο άρθρο, την πολιτική προστασία της συνθήκης Λισαβόνας. Όταν ξεκίνησε η Δανέζικη Προεδρία της διαπραγματεύσεις το Φεβρουάριο στην ομάδα εργασίας για μια νομοθετική πρόταση, μετά από τέσσερις μήνες ε, βλέπουμε που έχει φτάσει η πρόταση. Αποτιμούμε την όλη προσπάθεια που έγινε αυτούς τους τέσσερις μήνες. Νομίζουμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι για ένα συμβαστικό κείμενο. Η Κομισιόν είναι πιο έτοιμη στην ομάδα εργασία και για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα βασικά εκκρεμή θέματα. Με βάση αυτού του πρώτου απολογισμού που κάναμε ε, και αποτίμηση των απόψεων των κρατών μελών, μπορώ να σα πω ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν δισταγμού για τα νέα στοιχεία της πρότασης και τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες ακόμα για τις συνέπειες κάποιων από αυτά τα νέα στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη θεωρούν θετικό το ότι τώρα έχουμε αυτή την κωδικοποίηση. Τα δύο νομοθετήματα γίνονται ένα. Επίσης, τονίζω ότι τώρα αυτό η ευθυνική δηλαδή αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη ε, ξεκινάει από το μηδέν. Ήδη κάτι προβλέπεται, ήδη προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργασία σε διάφορου τομεί και ο στόχο είναι να έχουμε αλληλεγγύη προ τα κράτη-μέλη όταν τα χτυπά κάποια θεομηνία. Τα κράτη-μέλη επίση έχουν πει ότι θεωρούν θετικό το ότι είναι καλά δομημένη, διαρθρωμένη η καινούργια πρόταση για την πρόληψη και αντιμετώπιση γενικά των θεομηνιών. Επίσης κύριε Πρόεδρε σας ενημερώνω ότι η Δανέζικη Προεδρία αποφάσισε να γίνει μια συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο ε, Υπουργών Δικαιοσύνης τον ε, Ιούνιο, 8, 8 Ιουνίου ε, στο Λουξεμβούργο και ο στόχος της συζήτησης ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί έτσι τόσο ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Απλώς θα δώσουμε κατευθύνσει. θα επιταχύνουμε το ρυθμό των εργασιών και θα συζητήσουμε του τρει άξονε του, του, του θέματος που ακόμα βέβαια δεν μας έχουν βρει σύμφωνο στο ποιοι είναι ακριβώ αυτοί οι τρει άξονε. Πάντω, έχουμε κάποια καινούργια στοιχεία. Δηλαδή την ε, πρόταση όσον αφορά την χρηματοδότηση, τη συγχρηματοδότηση, τη μεταφορά το, το, την ομαδοποίηση των ενεργειών. Όλα αυτά πρόκειται να συζητήσουν οι Υπουργοί σε αυτή την συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη τον Ιούνιο. Οπότε, ε, συνοψίζω κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία του να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, τα νέα στοιχεία τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια συνένεση από τα κράτη-μέλη για κάποια ε, κοινή θέση. Και θα ενημερώσουμε φυσικά όταν πρέπει την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και τώρα. Κύριε Καρντίνη, η συγκήτρια. Ευχαριστώ. Τώρα. Ακούσαμε πολλούς συναδέλφους εξέφρασαν θετική άποψη. Τους ευχαριστώ γι' αυτό. Τους ευχαριστώ για την διάθεσή τους να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε αυτό το κείμενο που όπως είπε και η Κομισιόν και μου αρέσει αυτό που είπε η Κομισιόν είναι ένα εργαλείο που το θέλουν πολύ οι πολίτες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και το Συμβούλιο που θα συνέλθει τον Ιούνιο να ξεπεράσει τους όποιους δισταγμούς επί κάποιων σημείων. Γιατί πιστεύω ότι και οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες. Οι κυβερνήσεις χρειάζονται πολίτες που να θεωρούν αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στα θεσμικά όργανα της Βρυξέλλες ως ένα συνοθήλευμα από δράσεις που τους αφορούν. Ε, που θα θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό τους, στο πλευρό εκείνων που την έχουν ανάγκη. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω προς το παρόν, λοιπόν, τίποτα καινούριο. Σημειώνω αυτή τη θετική στάση και ελπίζω μετά από το Συμβούλιο του Ιουνίου να προκύψει η δυνατότητα για μία συμφωνία. Ελπίζω σε πρώτη ανάγνωση, δεδομένων και των προθεσμιών που έχουμε μέσα στο 2013. Ευχαριστώ κύριε Γκαρντίνη. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή θα ψηφίσει τις τροπολογίες 20 και 21 Ιουνίου προθεσμία για τις τροπολογίες 20-21 ναι, θα Προθεσμία για τις τροπολογίες ε, είναι 26 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα και θα γίνει μια συζήτηση των τροπολογιών 5 και 6 Νοεμβρίου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουμε 28 και 29 Νοεμβρίου και την Ολομέλεια του Ιανουαρίου του 2013 θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση και περνάμε στο επόμενο θέμα. Επαρθμόν 22. Προφορική ερώτηση του Chris Davis. Το θέμα είναι ζωολογική κήπη στην Ευρώπη. Ο Chris Davis έχει το λόγο για να κάνει το ερώτημά του. Thank you, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω είναι σωστό, αλλά έτσι όπως έχει τεθεί η ερώτηση, μήπως θα πρέπει πρώτα να δώσουν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν εγώ να συμπληρώσω. Κάνει μία αντίληψη λέει ο Πρόεδρος. Επομένω, τη σκητάλη έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Well, thank you very much, Chairman. And first of all, let me say that the European Commission... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη ικανοποίηση ε, ε διαπιστώνει ότι το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για ε, τους ευρωπαϊκούς ζωλίκους Κύπρος. Όσον αφορά τη σχετική οδηγία, θα γνωρίζετε ότι βασικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το να έχουμε κάποιο είδους βιώσιμη αηφόρο χρήση και αξιοποίηση της βιοπικιλότητος της άγριας ζωής με τα λεγόμενα in situ επιτόπια μέτρα. Και γι' αυτό και έχουμε και τις δύο σχετικές οδηγίες για τη φύση, αλλά έχουμε και τη σχετική στρατηγική για την βιοποικιλότητα που αφορούν και το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον, την υπόλοιπη υδρόγειο. Όμως, εδώ και κάποια χρόνια, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η οδηγία έχει ζωή υπέρ τη δεκαετία, αναγνωρίστηκε ότι θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την συντήρηση, την προστασία, γιατί θα πρέπει να τονιστεί ότι έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν ζωολογικοί κήποι εις την υπόθεση της βιοπικιλότητας. Και για αυτό πρόσφατα κάναμε μία μελέτη για αυτή την προστασία των ζωολογικών κήπων και με αυτή τη μελέτη στρατολογήσαμε τον ε, φορέα που συνενώνει τους ζωολογικούς κήπους της Ευρώπης. Ανεξάρτητο φορέα. Αναγνωρίζεται επομένω ότι όντω οι ζωολογικοί κήποι μπορούν να βοηθήσουν στον αφορά τη, τη βιοπικιλότητα, τη σωτηρία, την προστασία των ε, ειδών. Να, ο Λίγκας και το Μίνκ της Σιβηρίας και της Ευρώπης, αντίστοιχα. Και αυτό και έχει ρυθμιστεί, γιατί έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για αυτά τα δύο είδη. Οπότε και στο μέλλον πρόκειται να αναλάβουμε δράση και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Επίσης, Bon Free. Ε, έκανε άλλη μία σχετική μελέτη και έχουμε συνεχή επαφή αυτός ο φορέας επομένως έκανε έρευνα που προβληματιζόμαστε για το τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτές τις προσπάθειες του φορέα αυτού Γιατί δούλεψαν εις βάθος, ούτως ώστε να έχουμε επιχειρήματα να βασίσουμε τους ισχυρισμούς μας για την υπόθεση αυτή μια που είμαστε φύλακες των συνθήκων. Και έτσι θα αναλύσουμε τα δεδομένα για να δούμε αν χρειάζεται να ληφθεί δράση. Προς θέσπις νομοθεσίας πάντως, οι πρώτες επαφές με την Μπόμφρη μας κατέδειξαν ότι προτιμούν η Ευρωπαϊκή Επιστολή να μην, να μην νομοθετήσει καταρχήν. Και εκείνοι να μπορέσουν ε, να έχουν πιο δυναμικό ενεργό ρόλο για να έρθουν σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Εμείς ακολουθήσαμε τη συμβολή τους. Κάναμε αυτό το οποίο ζήτησαν και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων επαφών με τα κράτη-μέλη. Παρακαλώ. Πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι ο ρόλο μα είναι απλώ να πάλι θεύσουμε να διαπιστώσουμε αν γίνεται ορθή μεταφορά τη νομοθεσία και όντω τελικά είδαμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπω έπρεπε και γι' αυτό και ήδη, ήδη προσφύγαμε στο δικαστήριο το οποίο έλαβε κάποια πρώτη απόφαση οπότε το κράτος μέλος που δεν τα πήγαινε καλά με τη μεταφορά της νομοθεσίας τώρα έκανε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Και έτσι, θέλουμε να δούμε στη συνέχεια πώς θα καθοδηγήσουμε καλύτερα, πώς θα επιφέρουμε βελτίωση της διαχείρισης των ζωολογικών και πώς θα στρέψουμε τα κρατημέλη προς μια καλύτερη αξιοποίηση. Thank you very much. Now, Chris Davis, please. Thank you, Chairman. I very much welcome that. Ο Chris Davis, ευχαριστώ. Εκτιμώ την απάντηση της Κομισιόν. Χαίρομαι που ήρθε η Διευθύντρια να απαντήσει. Όπως ξέρουν οι βουλευτές, ε, εγώ ρώτησα γιατί ακριβώς δημοσίευσε τις εκθέσεις το Ίδρυμα, αυτό Born Free. Δεν μελέτησαν όλα τα κράτη-μέλη. Κατάλαβα πως επέλεξαν τυχαία ζωολογικούς κήπους, όμως η έκθεση φαίνεται πως είναι η συνολικότερη που έχουμε δει στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία. Δεν ξέρω αν έχετε δει την οδηγία, είναι συντομότατη. Ζητάει άδεια και προδιαγραφές ειδικά της προστασίας των ειδών και να προωθούν τη βιοπικιλότητα. Ζητάει να εκπαιδεύουν το κοινό και να φροντίζουν τα ζώα να κρατούνται σύμφωνα με τις ζωολογικές τους ανάγκες. Οι ζωολογικοί κήποι δεν είναι φυλακές, υποτίθεται είναι μέρη εκπαίδευσης και ευχαρίστηση Κανείς δεν θέλει να βλέπει τα ζώα να υποφέρουν. Νομίζω πως η έκθεση τονίζει το ότι πολύ συχνά δεν ε, πληρούνται οι προδιαγραφές, αλλά αυτό είναι ζήτημα άγνοιας ε, παρά κακίας. Μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ξεκινήσει διαδικασία σε παραβάση κατά όλων των κρατών μελών. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Καλό είναι να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, και να κινητοποιήσουμε την υιοθέτησή τους. Και υπάρχουν ζωολογικοί κήποι με υψηλά επίπεδα. Πολλά από αυτά είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ζωολογικών κήπων. 270 είναι στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχουν γύρω στις 4.000 ζωολογικοί κήποι. Οπωσδήποτε η ΆΖΑ, η Ένωση, έχει πολλή γνώση, αλλά είναι κρίμα ε, γιατί υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των οργανώσεων που ασχολούνται με τους ζωολογικούς κήπους. Π.χ. ο Λες Λιντίκη, ε, σοβαρός επαγγελματίας, ε, ε, απίθυνε μία επιστολή για να μην πάμε στην παρουσίαση του άλλου ιδρύματος, του Born Free. Γιατί αυτοί επίσημως δεν θεωρούν πως πρέπει να υπάρχουν ζωολογικοί κήποι. Αλλά τους έχουμε πει ότι θα υπάρχουν ζωολογικοί κήποι για κάναν αιώνα ακόμα, οπότε τουλάχιστον να είναι σε καλή κατάσταση. Ρεαλιστικό μου φαίνεται. Ίσως κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Ε, φέρτε τους εδώ πέρα να κάνουμε το σύμβουλο γάμου στην Επιτροπή μας μεταξύ των οργανώσεων αυτών. Συστάσεις τώρα για την Κομισιόν. Είπε η Διευθύντρια πως οι εκθέσεις αυτές ε, ε, βεβαίως ε, αντιμετώπισαν κάποια ζητήματα. Αναγνωρίζει η Κομισιόν πως το άρθρο 2 της οδηγίας είναι προβληματικό. Το άρθρο 2 λέει πως εάν οι ζωολογικοί κήποι δεν έχουν σοβαρό αριθμό ζώων μπορούν να εξαιρεθούν. Τι, και δεν ορίζεται ο σημαντικός αριθμός ζώων. Στην Ιταλία π.χ. υπάρχουν 60-70 ζωολογικοί κήποι και μόνο 8 έχουν άδεια. Δεύτερον, θα έρθετε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους για να απτυχθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς να βοηθήσετε τα κράτη μέλη να ερμηνεύσουν αυτή την οδηγία και να την εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά και αν γίνει αυτό πότε τρίτον θα κάνει η Κομισιόν περισσότερα για να συνεργαστούν οι επιθεωρητές των κρατών μελών μα <coughs> Ένα άτομο θα είναι σε κάθε χώρα. Για να συνεννοηθούν. Και τέλος, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας, αναφέρατε τη βιοπικιλότητα. Εάν όλοι οι ζωολογικοί κήποι που δεν έχουν άδεια, αλλά έχουν ζώα από απειλούμενα είδη, αν όλοι αυτοί συνεισέφεραν περισσότερο, τότε συλλογικά θα συνεισέφεραν όλοι οι ζωολογικοί κήποι. μπορείτε να κάνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ακούσαμε κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Τώρα είναι η κυρία Οκονή, ο Γιώ Λάινεν και Μπαριά κατόπιν. Παρακαλώ να είστε σύντομοι για να απαντήσει και η Κομισιόν σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Όμως το θέμα είναι σημαντικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε ρεαλιστές. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξή. Ότι μια ευρωπαϊκή οδηγία θε, θελήσανε να την ε, αξιοποιήσουν διάφορες ζωολογικοί κήποι πριν κάνετε τεθεί ισχύ μια που ακριβώς αφορά τα ενιδρία, αφορά τους σωλικούς κήπους. Όμως δεν εφαρμόζεται. Έχετε κάποιους ιδιοκτήτες ενιδρίων και ζωολογικών κήπων, οι οποίοι δεν είναι καλοί ιδιοκτήτες. Επίσης έχουμε κάποιους που κάνουν ανακαινήσεις, έχουμε κάποιους... Όπως όλες οι δουλειές, υπάρχουν καλοί και κακοί, εμπασίπτωση. Άρα, τι λύση έχουμε. Να νομοθετήσουμε εκ νέου και να θεσπίσουμε μια πιο σκληρή οδηγία. Αυτό το ζητούν πολύ, δεν το είπε ο κ. Ντέιβις. Έχουμε οδηγία. Ισχύει εδώ και 10 χρόνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμοθετήσουμε. Εξυπηρετεί τους σκοπούς μας. Και αυτό γιατί τι χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι ζωολογικοί κήποι και τα νηδρία. Και οι σωστοί έχουν μια χαρά εφαρμόσει αυτήν την οδηγία. Προστατεύει κάποια είδη, βοηθά στο να είναι σωστά η αναπαραγωγή των ζώων είναι ο πολλαπλασιασμός, ε, επίση επανεισαγωγή κάποιων ζώων, προστασία της βιοπικιλότητας, όλα αυτά τα πετυχαίνει η οδηγία. Άρα το έργο που τελείται είναι εξαιρετικό. Γιατί να ξανανομοθετήσουμε, γιατί να κάνουμε πιο σκληρή οδηγία και να ελπίσουμε ότι αυτοί που δεν εφήρμοσαν την πρώτη θα εφαρμόσουν τη δεύτερη. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, λέει αυτό το ίδρυμα που έκανε τη μελέτη να τους κλείσουμε αυτούς τους κακούς κήπους και να πάνε τα ζώα στην άγρια φύση. Αυτό δεν είναι λύση, γιατί οι ζωολογικοί κήποι προστατεύουν τη βιοπικιλότητα, προστατεύουν κάποια είδη. Είναι απαραίτητη η κήποι. Είναι φυσικά οικονομική δραστηριότητα, οπότε να μην έχουμε δογματισμούς για το περιβάλλον και να κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα αυτό που αφορά αυτή τη δραστηριότητα. Περίπου 3.500 θέσει εργασία 11.000 ε, έμεσα, δεκάδες χιλιάδες ε, σε όλη την Ευρώπη. Επομένω, υπάρχουν τα μέσα για την επίδευση των στόχων. Πρόκειται για μια προσθέμενη αξία. Πρόκειται για ε, τζίρο, πρόκειται για φόρου που πληρώνονται. Πρόκειται για μια κανονική οικονομική δραστηριότητα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τους κακούς να συμπεριφέρονται καλύτερα. Ευχαριστώ Γιολάινεν. Καλό είναι να συζητάμε για τους ζωολογικούς κήπους. Είναι πολύ σημαντική. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πάνε το χρόνο στους ζωολογικούς κήπους, πολλά παιδιά, νέοι, που μπορούν να μάθουν και τίποτα, αλλά πρέπει να είναι σωστές οι συνθήκες. Δεν χρειάζονται νέοι νόμοι, χρειάζεται εφαρμογή της υφισταμένης νομοθεσίας, όπως έλεγε και ο Οπότε θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή. Η επιτήρηση από την Κομισιόν, ε, συνεργασία των κρατών μελών, να μιλήσουν για προδιαγραφές, όλα αυτά τα ζητήματα της εφαρμογής. Θεωρώ πως δεν χρειάζεται τώρα ιδεολογικός αγώνας, ναι ή όχι, Υπάρχουν οι ζωολογικοί κήποι, έχουν καλές πτυχέ. Υπάρχουν ήδη που αλλιώ θα πέθαιναν. Επίση η εφαρμογή είναι το, το ζήτημα. Το α και το ω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλος. Άντερ Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Αντικαθιστώ την συνάδελφο, κυρία Άντερ Μπαρέα. Θεωρούμε ότι είναι ε, Τόσο στο συνάδελφο που αντικαθιστώ. Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση αυτή για τους ζωλικούς κήπους. Πρόκειται για επιχειρήσεις. Ε, προστατεύουν, φροντίζουν τα ζώα, ε, έχουμε εκεί μελέτες που γίνονται, τα προστατεύονται και ανέφερε ε, για τον Λίγκα της ε, Ιβηρίας και όχι της Ιβηρίας ε, οι Κομισιόν ότι έχουν σωθεί και αλλάζουν ρόλο. Και όχι, δεν πρόκειται περί έκθεσης επίδειξης των ζώων. Πρόκειται για, για, για επιμέλεια. Πρόκειται για προστασία που παρέχουν οι ζωολογικοί κήποι. Οπότε, στο άρθρο 2 έχουμε εδώ ένα παραθυράκι, ένα κενό σε σχέση με αυτήν την δεκαετή οδηγία η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί τόσο καιρό. Γιατί είπαμε τι γίνεται σε σχέση με την έγκριση, την άδεια. Ε, η άδεια ε, θεωρεί ότι και, και, και βεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, όσον αφορά τη λειτουργία. Άρα, αναδύονται δύο ερωτήματα. Πρώτα πρώτα, μας είπε η Κομισιόν να αλλάξουμε το άρθρο 2. Μας λέει για το άρθρο το προβλεπόμενο, όχι το προβλεπόμενο ποσοστό στο άρθρο 2 για να χορηγηθεί άδεια και έγκριση. Επίσης, μας είπε η Κομισιόν αλλά και άλλοι ότι δεν έχουν μεταφέρει στο ιστορικό δίκαιο όλα τα κρατημέρια την οδηγία. Ποιο είναι το ποσοστό των κακών μαθητών. Μην μου πείτε τα ονόματα. Πέστε μας το ποσοστό για να ξέρουμε πόσες είναι οι χώρες που μετέφεραν και που δεν μετέφεραν την οδηγία. Τελευταίο. Όσον αφορά ε, αυτό το φορέα που βοήθησε, εντάξει είναι εξωτερικός φορέας ε, και ενδιαφέρονται, εντάξει όπως συμβαίνει πολλές φορές. Όμως θα μπορούσαμε να έχουμε πιο αξιόπιστα δεδομένα μετά από κάποιους ελέγχους ε, αυστηρούς ε, η Κομισιόν τι, τι προβλέπει σχετικά. Ευχαριστώ. Τώρα ακούσουμε την Κομισιόν. Όσον αφορά βεβαίω τη χρησιμότητα των ζωολογικών κήπων ω πατέρας δύο κοριτσιών, θα συμφωνήσω με τον Γιολάινεν. Έχει, έχουν σημαντικό ρόλο. για να εξηγηθούν ε, και οι άνθρωποι με τα ζώα αυτά. Παρακαλώ λοιπόν, απαντήστε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, η πρώτη ερώτηση που έκανε ο Κρίς να την απαντήσω. Έχουμε πρόθεση, χάρη σε, αυτά τα νέα, σε αυτές τις νέες συμβάσεις που ετοιμάζουμε να βοηθηθούμε από έναν εξωτερικό ε, εταίρο, ούτως ώστε να ετοιμάσουμε αυτά τα έγγραφα καθοδήγησης. Θα σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους, με το Born Free Association, με άλλες οργανώσεις, με τα κράτη-μέλη φυσικά, γιατί φυσικά τα κράτη-μέλη είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι για τους ζωολογικούς κήπους και με τους επιστήμονες. Μην ξεχνάμε ότι η ουσία που μας απασχολεί, που είναι να έχουμε καλό επίπεδο διατήρησης και να προστατεύσουμε τα είδη ζώων, είναι σημαντικό να έχουμε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια και τους ε, επιστήμονες. Δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στο τέλος πάντως θα ε, συγκαλέσουμε μια συνάντηση με όλους τους ενδιαφέρομενου φορείς και με τα κράτη-μέλη και θα υποβάλουμε στα κράτη-μέλη το αποτέλεσμα της δουλειά αυτής. Και ελπίζουμε να πάρουμε τη δέσμευση από τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν από εκεί και πέρα. Αυτό είναι το πρώτο. Επίσης, άλλε παρεμβάσει ζήτησαν να του πούμε τι κάνουμε στην πράξη. Μαζί με τους συναδέλφους που ασχολούνται με την υγεία, κάνουμε ε, σεμινάρια κατάρτισης για κτηνίατρους που δουλεύουν σε ζωολογικούς κήπους στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να αφυπνιστούν Ω προ τι ανάγκε για καλύτερη προστασία και συντήρηση και διατήρηση των ειδών στους ζωολογικού κήπου. Για το άρθρο 2 τη οδηγία. είναι και για τη σημασία του όρου significant ο Chris Davis ε, έχει αρκετή εμπειρία και έχει συμμετάσχει, έχει συνεισφέρει όπως και πολλοί από εσά, σε πολλές νομοθετικές διαδικασίες. Και αναγνωρίζω ότι η σαφής νομική σύνταξη δεν είναι πάντα το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Θα προσπαθήσουμε βέβαια το οποιοδήποτε νομοθέτημα υποβάλλουμε να είναι και εύληπτο και εύκολο στην εφαρμογή. Τώρα για αυτό το θέμα του σημαντικού, του significant. Ξέρετε ότι και σε άλλα νομοθετήματα έχουμε τις ίδιες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο, κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε μια ερμηνεία. some other questions. Να έρθω τώρα σε κάποια άλλα ερωτήματα. Δύο συγκεκριμένα. Από το είναι το ένα για τις επιθεωρήσεις της Κομισιόν. Ο πρώτος θεματοφύλακας της νομοθεσίας είναι τα κράτη-μέλη. Και καταρχήν τα κράτη-μέλη πρέπει να διενεργήσουν τις σωστές επιθεωρήσεις. Όπως θα ξέρει η Επιτροπή σας Περιβάλλοντος, η Κομισιόν ε, θέλει να αναθεωρήσει μια σύσταση για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Υπάρχει ήδη μια σύσταση αφορά περιβαλλοντικά θέματα, νομοθεσίες περιβάλλοντος, αλλά με περιεχόμενο βιομηχανικό. Δεν αφορά σχετική νομοθεσία με περιεχόμενο διατήρησης ειδών. Δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσουμε, θα εξετάσουμε και τέτοια θέματα διατήρησης ειδών, και τα λοιπά και της φύσης. Γιατί αυτή είναι μια μακρόπνοη προσπάθεια που μπορεί να μας πάει πολύ μακριά. Τώρα, ένα θέμα ότι δεν έχουν μεταφέρει όλα τα κράτη-μέλη πολύ σωστά την ε, σχετική νομοθεσία. Ίσως με παρερμηνεύσατε, Πρόεδρε. Συγγνώμη. Η μεταφορά της οδηγίας έγινε σωστά στα κρατημέλη. Μόνο μία περίπτωση έχουμε όπου φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Το εν λόγω κρατός μέλος διόρθωσε την εθνική νομοθεσία μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επομένως έχουμε πλήρη και σωστή μεταφορά της ε, οδηγίας. Ευχαριστώ τις δηλώσεις και τις απαντήσεις της Κομισιόν. Τώρα να ευχηθώ καλή όρεξη και τα λέμε 3 η ώρα. Το έχουμε την Κόνη Χέντεγκάρτ εδώ πέρα. Παρακαλώ να είστε λοιπόν στην ώρα σας. Γεια σας.